Sinon, je voulais vous dire que ce matin, nous avons désigné un rapporteur. Να σα πω ότι σήμερα το πρωί ορίσαμε ένα εισηγητή για το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο. Και μια και δεν υπάρχει άλλο εισηγητή, θα το αναλάβω εγώ. Ε, είναι ένα πραγματικά σημαντικό σημείο. Σας ευχαριστώ που δεν ζητήσατε κάποιοι ε, να γίνετε εισηγητές. Προφανώ ήταν όμως και κάτι το απρόβλεπτο επί της δημοσιονομικής διαδικασίας για το 2016. Ορίσαμε για εισηγητή για τους υπόλοιπους τομείς και κλάδους τον κύριο Ντεπρέ, τον Ζεράρ Ντεπρέ. Η Επιτροπή Προϋπολογισμών θα προετοιμάσει μία γνωμοδότηση για το λεγόμενο Green Growth Opportunities, ευκαιρίες πράσινης ανάπτυξης. Όλοι συνειδητοποιούν το δυναμικό που παρουσιάζουν τα θέματα της ενέργειας, της ενεργειακής μετάβασης και της πράσινης ενέργειας. Ο εισηγητής θα οριστεί ε, σύντομος. Εφόσον κάποιος ενδιαφέρεται μπορεί να καταθέσει και την υποψηφιότητά του όπως γίνεται συνήθως. Ταυτόχρονα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πάρει μέρος στην λεγόμενη Ευρωπαϊκή Κοινοβουλευτική Εβδομάδα μέσω της εφαρμογής του άρθρου 13 της συνθήκης Fiscal Compact. Θα πρέπει εμείς να εκφράσουμε τις επιθυμίες τις οποίες θα θέλαμε να δούμε να συζητώνται, να αντιμετωπίζονται στα πλαίσια αυτής της συνάντησης θα υπάρξουν αντιπροσωπείες από πλευρά των κοινοβουλίων της ζώνης ευρώ και έχουμε την ευκαιρία να στείλουμε ένα ισχυρό μήνυμα γύρω από το θέμα των απλήρωτων λογαριασμών. Με αυτόν τον τρόπο νομίζω ότι θα μπορέσουμε να ευαισθητοποιήσουμε τα κοινοβούλια των κρατών μελών. Γιατί τα χρέη της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι χρέη των κρατών μελών. Γύρω από το θέμα των μελετών επικυρώσαμε τις προτάσεις τις οποίες έκαναν ε, οι συνάδελφοι της Επιτροπής Προϋπολογισμών για την παραγωγή των ιδίων πόρων και για την σύσταση των ομάδων των εμπειρογνωμόνων. Αυτά είναι αιτήματα τα οποία καταθέτουμε σε συνεργασία με τους συναδέλφους της Επιτροπής Ελέγχου Προϋπολογισμών. Τώρα, για τους εμπειρογνώμονες σε συνεργασία με την Επιτροπή Ασφάλειας και Άμυνας. Θα ζητήσουμε την άδεια να μιλήσουμε για την αμοιβεοποίηση ορισμένων εξωτερικών υπηρεσιών. Ίσως τα κράτη-μέλη θα μπορούσαν εδώ να βρούνε κάποιους ε, χώρους εξοικονόμησης χρημάτων, μιλώντας, παράδειγμα είναι αυτό, για κοινέ πρεσβείες ανάμεσα στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε σε ποιο επίπεδο μπορούμε να εξοικονομήσουμε χρήματα και σε εθνικό επίπεδο, ακριβώς μέσω του συνδυασμού χρήσης μέσων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Εφόσον μπορείτε να μας δώσετε ονόματα εμπειρογνωμόνων γύρω από όλα αυτά, είμαι στη διάθεσή σας. Θα τα σημειώσουμε. Δεν έχω άλλες ε, ανακοινώσεις να κάνω από πλευράς Προεδρίου στην αρχή της συνεδρίασης. Περνάμε τώρα στο... στην κατάληξη των ε, διαπραγματεύσεων με το Συμβούλιο, την αποτυχία του... της συνδιαλλαγής και την επίτευξη μιας συμφωνίας στον τριγωνικό διάλογο μια συμφωνία η οποία έχει συγκεκριμενοποιηθεί τη Δευτέρα το βράδυ. Να ευχαριστήσω καταρχήν όλους αυτούς οι οποίοι έλαβαν μέρος στην διαδικασία αυτή, τα μέλη της Επιτροπής μας. Μπορέσαμε να προχωρήσουμε τόσο πολύ γιατί υπήρξε ενότητα μαζί μας. Και σας ευχαριστώ για αυτό. Ευχαριστώ φυσικά και τον τους εισηγητές οι οποίοι ήταν μονίμως παρόντες στις συνεδριάσεις αυτές συνέβαλαν στην εκπόνηση της κοινή δήλωσης και οι οποίοι έπαιξαν σημαντικό ρόλο στο να μπορέσουν οι διαπραγματεύσεις αυτές να ξεπεράσουν το στάδιο της ματέωσης. Και φυσικά στρέφομαι προς τους ε, εισηγητές, τις εισηγήτριες ίσως καλύτερα, όταν κάποιο αποφασίζει να είναι μέλος τη Επιτροπής των Προπολογισμών, έχει να λάβει πολύ σημαντικές αποφάσεις. Και ο δρόμος που πρέπει να ακολουθήσει είναι σκολιός και γεμάτος ματαιώσεις και αυταπαρνήσεις. Αλλά γυναίκες και άνδρες πολιτικοί που θέλετε να εξασφαλίσετε την ε, επικράτηση της αλήθειας και όχι το να αποστρέφει κανείς το πρόσωπό του από την πραγματικότητα. Γι' αυτό θέλω να σας αποτίσω φόρο τιμής. Το αποτέλεσμα βέβαια δεν ήταν αυτό το οποίο προσδοκούσαμε. Έχουμε επιτύχει να βελτιώσουμε το επίπεδο των πιστώσεων πληρωμών κατά 4,8 δισεκατομμύρια ευρώ εκεί που περιμέναμε για το 2014-2015 7 δισεκατομμύρια. Γιατί σύντομα αρχίζει το έτος 2015, ότι δεν πληρωθεί το 2014 θα πρέπει να πληρωθεί το 2015. Ζητήσαμε 7 και πήραμε στην πράξη 4,8 δισεκατομμύρια ευρώ. Σε ό,τι αφορά τις πιστώσεις υποχρεώσεων, δείξαμε μεγάλη αυταπάρνηση εδώ και εδώ Υπήρξε εξαίρετο έργο από τον Γενικό Εισηγητή του Προϋπολογισμού, αλλά φαντάζομαι ότι αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να οδηγήσει σε μεγάλη απογοήτευση. Παρ' όλα αυτά, πιστεύω ότι τους επόμενους μήνες και τα επόμενα χρόνια θα αποδώσουν καρπούς αυτές οι προσπάθειές μας. Με τα 4,8 δισεκατομμύρια δεν έχουμε καν καταφέρει να σταθεροποιήσουμε τα ραλ, τα ποσά προς εκταμίευση που δεν έχουν πληρωθεί. Και δεν μπορούμε λοιπόν να πούμε ότι μπαίνουμε καν σε μια διαδικασία εκαθάρισης αυτών των ποσών. Κάτι το οποίο ζητήσαμε από την Κομισιόν να εξασφαλίσει μαζί με τα άλλα θεσμικά όργανα. Θέλουμε από την Κομισιόν να μας πει ποιο είναι το επίπεδο το οποίο μπορεί να θεωρηθεί αποδεκτό για αυτά τα μη πληρωμένα, ποσά που δεν έχουν πληρωθεί, ίσως 10 δισεκατομμύρια, η Κομισιόν θα πρέπει να μας πει ποια είναι τα ποσά που δεν θα έχουν πληρωθεί στις 31 Δεκεμβρίου 2014 και επομένως την απόκληση ανάμεσα στο, στην πραγματικότητα και στο στόχο του να μην ξεπεράσουμε πραγματικά τα 10 δισεκατομμύρια και όλα αυτά πρέπει να αποτελέσουν το αντικείμενο ενός σχεδίου εκαθάρισης των υπολείπων. Πρέπει να συνεχίσουμε την πίεσή μας στους επόμενους μήνες τόσο προς την Κομισιόν όσο και προς το Συμβούλιο. Εγώ με τον κύριο Ταράντι ήμουνα στην κοινή συνεδρίαση Επιτροπή Προπολογισμών, Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων και φυσικά αναφερθήκαμε στο θέμα των πληρωμών. Το μνήσαμε ότι όλο το 2014 είχαμε να αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα, αυτό το όνειρο. Δηλαδή, ήμασταν ιδιαίτερα φιλόδοξοι ό,τι αφορά τη χρηματοδότηση τη Ουκρανία, χωρί όμω να υπάρξει η απαραίτητη ρύθμιση σε επίπεδο πληρωμών. Μα εξήγησε ο εκπρόσωπο του Συμβουλίου, οι υποχρεώσει είναι εύκολε. Μόνο για τι πληρωμέ έχουμε δυσκολία όταν πρέπει να πληρώσουμε. Και μα είπε ότι υπάρχουν όλοι αυτοί οι λογαριασμοί στον τομέα των εξωτερικών υποθέσεων που θα πληρωθούν μόνο το 2015 αντί το 2014. Για όλα αυτά λοιπόν ζητώ από εσά να μην αφήσετε το Συμβούλιο να ξεφύγει από τι υποχρεώσει του και να ασκήσετε πίεση σε εθνικό επίπεδο, να μιλήσετε στους συναδέλφους σας των ε, βουλών και των γερουσιών στο εθνικό επίπεδο και να τους εξηγήσετε ότι υπάρχει ένα πάρα πολύ σοβαρό πρόβλημα το οποίο δεν μπορούμε να παραγνωρίσουμε, το πρόβλημα των λογαριασμών που ακόμα δεν έχουν εξοφληθεί. Υπάρχει επίσης και η ιδέα που ανέφερε ο κ. Φερνάντης ότι στη βδομάδα που συναντάμε τα Εθνικά Κοινοβούλια να εξασφαλίσουμε την συζήτηση αυτού του σημείου όταν θα είναι παρόντες και οι συναδελφοί μας από τα Εθνικά Κοινοβούλια. Αυτά λοιπόν και για τα ειδικά μέσα. Υπάρχει μια κοινή δήλωση όπου αναφέρεται η άποψη του Συμβουλίου αλλά και του Κοινοβουλίου σε χωριστές ουσιαστικά κοινέ δηλώσεις και αναφέρεται, μπορεί να δει κανείς από αυτές τις δύο δηλώσεις, πόσο μεγάλη είναι η απόσταση που μας χωρίζει από το Συμβούλιο και τώρα μπορώ να δώσω το λόγο στους συζητητές μας και ξεκινώ με την κυρία Γκουάρδα Σαραλ. <coughs> Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Πολλές φορές συζητήσαμε το θέμα αυτό στην Επιτροπή μας και μας αναφέρατε ήδη πώς πήγαν οι διαπραγματεύσεις ή μάλλον πώς δεν πήγανε, πώς δεν προχωρήσαν οι διαπραγματεύσεις. Απλώς αυτό είναι το, η τελική απόλυξη μιας διαδικασίας που ήταν πάρα πολύ δύσκολη για μας και για το Κοινοβούλιο, αλλά φυσικά η κάθε, κάθε θεσμικό όργανο επέχει τη δικιά του ευθύνη και είναι υπεύθυνο για τη δική του εργασία. Ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη και εργόδης και σκληρή διαδικασία και για τα τρία θεσμικά όργανα, τα οποία ενεπλάχισαν στις διαπραγματεύσεις για τον προϋπολογισμό. Για το αποτέλεσμα Τώρα μπορεί να δει κανεί το ποτήρι μισογεμάτο ή μισοάδιο. Εμείς είχαμε προσδοκίες πιο ψηλές βέβαια. Ο στόχος μας ήταν, το είχαμε πει από την αρχή και ήταν κάτι που ερχόταν από την προηγούμενη εντολή μας, ο στόχος μας ήταν να προσπαθήσουμε να λύσουμε το πρόβλημα των μη εξοφλημένων λογαριασμών ή τουλάχιστον να υπάρξει κάποιο, <clears throat> κάποια οδός ομαλής προσγείωσης για αυτά τα ποσά Θέλαμε να δούμε αν αυτές οι διαπραγματεύσεις και όλα αυτά τα οποία είχαμε υπογράψει σε κοινή δήλωση των τριών θεσμικών οργάνων θα μπορούσαν να γίνουν πραγματικότητα ή όχι. Για τα αριθμητικά στοιχεία και πάλι μπορεί κανείς να έχει διαφορετικές αναγνώσεις. Είναι σαν τις εκλογές που όλοι κερδίζουν και κανείς δεν χάνει. Αν θέλουμε να τα δούμε θετικά τα πράγματα μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Αν λάβουμε υπόψη την αντίδραση του Συμβουλίου σε οποιαδήποτε αύξηση ακόμα και για ένα ευρώ, το γεγονός ότι καταφέραμε να εξασφαλίσουμε τα 4,87 ε, δισεκατομμύρια ευρώ είναι μια κάποια επιτυχία. Σε κάθε συνάντηση με το Συμβούλιο καταφέραμε να κερδίσουμε και λίγο περισσότερο και να αποσπούμε λίγο περισσότερο από το Συμβούλιο. Δεν ήταν εύκολο. Δυστυχώς <clears throat> δεν μπορέσαμε να συζητήσουμε αρκετά τα θέματα αυτά των περικοπών που έχει επιφέρει το Συμβούλιο σε πολλές κατηγορίες του προπολογισμού που για μας είναι πάρα πολύ σημαντικές. Εμείς εξασφαλίσαμε να μην γίνουν αυτές οι περικοπές και σε ορισμένες περιπτώσεις να πετύχαμε και ορισμένες μικρές αυξήσεις οι οποίες έχουν μάλλον συμβολικό χαρακτήρα αλλά έχουν σημασία για τις ε, ε, θέσεις αυτές του προϋπολογισμού. 12 εκατομμύρια σε, σε σύνολο 140 εκατομμυρίων είναι αρκετά λεφτά και κυρίω γιατί προορίζονται αυτά τα ποσά για τις υποτροφίες του Εράσμους που έχει μεγάλη συμβολική σημασία για την Ευρώπη 10 εκατομμύρια παραπάνω για την ανθρωπιστική βοήθεια ή 22 εκατομμύρια παραπάνω για να βοηθήσουμε τα 5 εκατομμύρια ε, προσφύγων στη Μέση Ανατολή. Όλα αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά. Προφανώς λένε δηλαδή, είναι αυτό το οποίο ήθελε το Κοινοβούλιο, θέλαμε πολύ περισσότερα. Αλλά την Δευτέρα το βράδυ, όταν έπρεπε να καταλήξουμε ή όχι σε μια συμφωνία, θεωρήσαμε ότι δεν μπορούσαμε να προχωρήσουμε περισσότερο, δεν μπορούσαμε να αποσπάσουμε περισσότερο από το Συμβούλιο και μια ρήξη στις διαπραγματεύσεις δεν θα βοηθούσε καθόλου ούτε εμά ούτε την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν μπορούσαμε να πετύχουμε πολύ περισσότερο. Και το Συμβούλιο είχε φτάσει και αυτό με τις παραχωρήσεις σε ένα σημείο το οποίο δεν μπορούσε να υπερβεί. Δεν ξέρουμε λοιπόν τι θα είχε γίνει αν θα ήταν καλύτερα να υπάρξει μια ρίξει και μια διακοπή των διαπραγματεύσεων. Εμείς κρίναμε ότι ήταν καλύτερο να δεχτούμε αυτό το οποίο μπορούσαμε να επιτύχουμε και περιμένουμε φυσικά και το σχέδιο Juncker. Ελπίζουμε ότι με την εφαρμογή αυτού του προπολογισμού μπορούμε να, να ξεκινήσουμε και τη διαπραγματεύση για το <coughs> σχέδιο αυτό Juncker. Ήταν λοιπόν γλυκό πικρό το αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων. Κάποια πράγματα πήγαν καλά, κάποια όχι και τόσο. Το 2015 θα έχουμε την ευκαιρία να κάνουμε μια πιο γαλήνια αποτίμηση αυτών των διαπραγματεύσεων και ελπίζω ότι με την βοήθεια των ε, επομένων προεδριών από την 1η Ιανουαρίου θα μπορέσουμε πια να εργαστούμε για να μειώσουμε τα υπόλοιπα προσπληρωμή <coughs> τα οποία εκκρεμούν Περιμένουμε από την Κομισιόν να μας παρουσιάσει προτάσεις και περιμένουμε και από τις δύο επικείμενες προεδρίες του Συμβουλίου να συμβάλλουν σε κάτι τέτοιο. Επομένως να μπορέσουμε έτσι να θέσουμε ένα τέρμα σε αυτήν την πολύ δυσάρεστη κατάσταση για τα προσεκταμίευση ποσά που δεν έχουν πληρωθεί. Θέλω πριν κλείσω να ευχαριστήσω και τον Πρόεδρό μας για την προσπάθεια που κατέβαλε, αλλά κυρίως τη Γραμματεία, η οποία έκανε μια καταπληκτική, μια ε, τεράστια προσπάθεια για τις τροπολογίες, για την αξιολόγηση των προτάσεων του Συμβουλίου. <clears throat> Εργάστηκαν με τρομερή πίεση, αναγκάζοντας να αντιμετωπίσουν με ένα οριμαγδό από αριθμούς και προσπαθώντας να εξασφαλίσουν ότι δεν θα υπήρχαν αριθμητικά λάθη. Λοιπόν, θέλω να αποτίσω φόρο τιμή στη Γραμματεία για το έργο της και τη βοήθεια που μας προσέφερε. Πρόεδρε, συνάδελφοι, σε άλλες καταστάσεις τα πράγματα ήταν λίγο πιο απλά από τη συγκεκριμένη περίπτωση που προσπαθήσαμε από καινού να πετύχουμε ό,τι καλύτερο γίνεται σε άλλα θεσμικά όργανα. Τα πράγματα φαίνεται ότι είναι καλά. Το Συμβούλιο αναγνώρισε ε, ότι χρειάζεται να εξαγάγουμε συμπεράσματα από την απόφαση του δικαστηρίου και ότι θα πρέπει να κοιτάξουμε τι θα γίνει με τις ε, οικονομικές απαιτήσει και με το κείμενο και κατά δεύτερον σε ό,τι αφορά την εξωτερική υπηρεσία, την υπηρεσία εξωτερικής δράσης και το σχετικό κόστος προκειμένου να διαμορφωθεί με λειτουργικό και αποτελεσματικό τρόπο το όργανο αυτό και να μην ε, κατακαιρματίζεται το έργο της, να μην υπάρχουν πέντε γενικές διευθύνσεις και 15 ε, διαφορετικές γραμμές του προπολογισμού και τελικά όλα να καθυστερούν. Αυτό είναι θετικό βήμα και κατά τρίτον πετύχαμε στη συνεργασία ως Κοινοβούλιο με την Επιτροπή των Επιτροπών, αλλά και με την Επιτροπή, την Οικονομική και την Κοινωνική, να κάνουμε ένα πρώτο βήμα στη συνεργασία Και από τις δύο λοιπόν επιτροπές πήραμε υπαλλήλου προκειμένου να οικοδομήσουμε μια κοινή ε, επιστημονική ε, διεύθυνση. Δεν ήταν τόσο σύμφωνο το Συμβούλιο, εμείς ε, παρόλα αυτά το δηλώσαμε πολύ απλά, ήταν καλό βήμα. Στην αρχή υπήρχε και μια παρανόηση, δυστυχώ από δική μας πλευράς και αυτό σήμαινε ότι πρέπει να γίνουν συζητήσεις σε διαφορά μείωση 5% του προσωπικού γιατί αυτό προέκυψε από μία παρανόηση σε ένα πίνακα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε ό,τι αφορά τη συνεργασία, τις διαφορές που προκύπτουν από την εσωτερικοποίηση και την εξωτερικοποίηση και εμείς δεν τα είχαμε συμπεριλάβει, το Συμβούλιο τα είχε συμπεριλάβει. Απορρίψαμε λοιπόν τον πίνακα αυτό μετά από συζητήσεις με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στη τελική ανάλυση διαγράφηκε όλη η Επιτροπή γιατί αυτό θα σήμαινε ότι δεν θέλουμε επιπρόσθετο προσωπικό για τις ε, οργανισμού. οργανισμούς γενικότερα. Ε, αυτό δεν μας έβρισκε σύμφωνος και γι' αυτό λοιπόν καταρκήσαμε και διαγράψαμε όλη την παράγραφο και αυτό απλοποίησε τα πράγματα. Σε ό,τι αφορά τον γενικό προϋπολογισμό θα ήθελα να πω δύο-τρεις κουβέντες μόνο. Θεωρώ ότι ήταν σημαντικό το ότι προσπαθήσαμε να συνεχίσουμε χωρίς ε, διαλύματα της διαπραγματεύσεις και χωρίς όμως να κάνουμε έκπτωση στην αρχή του ότι πρέπει να πληρώνονται πάντα οι παλιοί λογαριασμοί. Και νομίζω ότι καταφέραμε να μαζέψουμε και να συλλέξουμε κάπως το σεβασμό του Συμβουλίου. Δεν ήταν θέμα συζήτησης, ήταν θέμα μόνο του το, το, το ότι πρέπει να τηρούνται οι συνθήκες. Δεν είναι δυνατόν νέα καινούργια προγράμματα να μην ξεκινάνε και από αυτά τα χρήματα να πληρώνονται οι παλιοί Και αυτό που με φαίνεται πάρα πολύ ενδιαφέρον είναι το σχέδιο πληρωμών. Συνήθως το Συμβούλιο είναι αυτό που λέει ότι θα πρέπει να είμαστε συνεπείς και διαφανείς. Αλλά όταν ζητήσαμε εμείς ένα κείμενο για τη συνέπεια αυτή των πληρωμών, έκανε πίσω και το Συμβούλιο για τεχνοκρατικούς λόγους και με τεχνοκρατικές ε, δικαιολογίες. Και πραγματικά θαυμάζω και τον Ζεράρ και τον ε, Πρόεδρο και τους άλλους δύο εισηγητές που συνέχισαν να απαιτούν τα συμφωνημένα. Θα πρέπει λοιπόν να καλέσουμε και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά και να αναγκάσουμε το Συμβούλιο να επιβάλλουν διαφάνεια σε ό,τι αφορά τις πληρωμές παλαιών προγραμμάτων και των ε, καινούριων προγραμμάτων, προκειμένου να τα συζητούν αυτά μαζί μας. Να μην βρισκόμαστε πάντα σε μια γκρίζα ζώνη που τελικά ούτε εμείς οι ίδιοι δεν ξέρουμε τι συμβαίνει ακριβώς. Γι' αυτό λοιπόν πιστεύω ότι είναι καλό και πραγματικά θα πρέπει να ακολουθήσουμε αυτή την τακτική τους επόμενους μήνες. Αυτό θεωρώ ότι είναι η μεγάλη επιτυχία του ότι περάσαμε με στέλνους <clears throat> αυτή την στάση. Σας ευχαριστώ. το Ευχαριστώ πρόεδρε. Όπως και οι δύο προλαλήσαντες θέλω να ευχαριστήσω το σύνολο των μελών της Επιτροπής και τη Γραμματεία. Μπορέσαμε να διαπραγματευτούμε διότι γνωρίζαμε ότι υπήρχε μια κάποια συνένεση και είναι πολύ πιο εύκολο να διαπραγματεύεται κανείς όταν ξέρει ότι πίσω του υπάρχει ομοφωνία. Θέλω να ευχαριστήσω και εσάς κύριε Αρτουρή γιατί εμείνατε στη γραμμή μας και αποδείξατε την αποφασιστικότητά μας, η οποία αμφισβητήθηκε. Ευχαριστώ τη Γραμματεία και τους συνεργάτες μας. Και να ευχαριστήσω ιδιαιτέρως ε, την ε, κυρία Γουάρδια Ζάμπαλ... την Άιντερ, γιατί αυτή στιγμή ε, έδειξε ότι είναι αλληλέγγυη με τις θέσεις μας για τις πληρωμές του 2014 τότε ε, τα περιθώρια για το 2015 είχαν αρχίσει να μικραίνουν και είδα εκεί τις ικανότητές της και την επίδειξη αλληλεγγύης την οποία έκανε απέναντι στις θέσεις μας. Θα ήθελα να μου επιτρέψετε εδώ να μιλήσω λίγο άσχημα, θα το πω δηλαδή κάπως απότομα. Ευτυχώς που τέλειωσε αυτή η ιστορία γιατί κάθε φορά που κατέβαινε μια νέα πρόταση και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκανε μια συμβιβαστική πρόταση ήταν τρεις χειρότερη από την προηγούμενη. Ξέρω ότι δεν αρέσει αυτό που λέω αλλά καλό είναι που ξεμπερδέψαμε. Καλά κάνετε, είναι ανακουφιστικό που το λέτε λέει ο πρόεδρος γιατί αλλιώς ε, θα μας ε, έπαιρναν τα εσώρουχα σε εισαγωγικά και το θέαμα θα ήταν όπως φαντάζεστε ιδιαίτερα δυσάρεστο λέει ο κ. Ντεπρέ. Από την άλλη η απογοήτευση δεν συνιστά πολιτική θέση. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε και τι θετικά στοιχεία υπάρχουν. Εγώ έκανα κάποιους μικρούς υπολογισμού για το 2014. Εμείς ζητούσαμε συνολικά 4 δις 700 φρέσκο χρήμα. Τώρα τι έχουμε. 3 δις ε, 29 εκατομμύρια, δηλαδή είμαστε γύρω στο 60% από αυτό που ζητούσαμε. Τι μας έδινε το Συμβούλιο στην αρχή, μηδέν, τίποτα. Δηλαδή πήραμε το 68% αυτού που ζητάγαμε. Και αν προσθέσουμε εδώ και κάποιες επιμέρους ε, μεταφορές έχουμε 4.200 με τις αναδιατάξεις, με τις αναβολές πρωτοβουλειών. Υπάρχουν λοιπόν για το 14 4 δις 200 εκατομμυρία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν εκεί όπου απαιτούνται ταχύτατα πληρωμές. Είναι φυσιολογικό λοιπόν να είμαστε απογοητευμένοι γιατί δεν πετύχαμε το σύνολο των στόχων μας. Από την άλλη όμως δεν θα πρέπει να πούμε ότι στα πλαίσια μιας διελκυστίνδας εμείς ιτηθήκαμε. Όχι. Αντικειμενικά μπορούμε να πούμε βλέποντας τα αποτελέσματα της διαπραγμάτευσης ότι εμείς βγήκαμε νικητές από τη διαδικασία. Το θέμα είναι τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Να δούμε δηλαδή το λειτουργικό πρόγραμμα απορρόφησης των χρεών, το οποίο εσείς και αγραφήσατε λίγο πρόεδρε. Θα πρέπει να συμφωνήσουμε με το Συμβούλιο γι' αυτό. Το Συμβούλιο δεν ήθελε να βάλουμε τη φράση στα αγγλικά «will agree». Όχι, ήθελε μια φράση που έλεγε «κοιτάξτε θα προσπαθήσουμε μήπως και...» Όχι, τώρα έχουμε δεσμεύσει τουλάχιστον σε επίπεδο αρχή στο Συμβούλιο. Και νομίζω αρχη το συμβουλιο και νομιζω οτι τον επόμενο χρόνο θα μπορέσουμε κρατώντας τον προσανατολισμό μας να προχωρήσουμε στο σχέδιο απορρόφησης των απλήρωτων λογαριασμών, των χρεών μας και αυτό έχει ουσία. Και αν μείνουμε ενωμένοι όπως σήμερα έχουμε πολλές ελπίδες να κερδίσουμε. Ευχαριστώ κύριε Ντεπρέ. Πράγματι, αν είχαμε καταλήξει στην πλήρη αποτυχία. Τότε στην περίπτωση αυτή τα 5 δισεκατομμύρια πόρων του 2014 που προέρχονται από τα πρόστιμα που επευλήθηκαν δεν θα ήταν κομμάτι των πιστώσεων πληρωμών. Αυτό λοιπόν το περίσσευμα της, ε, του οικονομικού έτους 2014 θα ξαναγίζει στα θησαυροφυλάκια των κρατών μελών. Είναι και αυτό το επιχείρημα λοιπόν, το οποίο τόνισε ο κύριος Δεπρέ κατά τις διαπραγματεύσεις. Είναι ένα πολύ ισχυρό επιχείρημα. Στο μέλλον θα θέλαμε η θέση της Κομισιόν να είναι σταθεροποιημένες. Κύριε Φερνάντης. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρο και εγώ θέλω να συγχαρώ όλους αυτούς οι οποίοι έλαβαν το λόγο προηγουμένως και φυσικά συνέβαλαν στις διαπραγματεύσεις. Πρώτα απ' όλα στον πρόεδρο της Επιτροπής μας για τον τρόπο που διεξέχθησαν διαπραγματεύσεις, στους εισηγητές, στις πολιτικές ομάδες, στη γραμματεία που έκανε πολύ μεγάλη δουλειά, στα πολιτικές ομάδες που έπαιξαν σημαντικό ρόλο που ήταν πολλές φορές αόρατος. Νομίζω ότι μπορούμε να είμαστε ικανοποιημένοι για την καλή εργασία που κάναμε. Όσοι έχουν διαφορετική άποψη, νομίζω ότι θα πρέπει να ξέρουν ότι θα ήταν αδύνατο να δικαιολογήσουμε ενώπιον της κοινή γνώμης την απόρριψη μιας συμφωνίας. Βάλαμε το Συμβούλιο στο σωστό δρόμο δεν ήθελε το Συμβούλιο να χρησιμοποιήσει τίποτα από τα ποσά που ήταν διαθέσιμα για να πληρώσει τα, τους λογαριασμούς που ήταν προς εξόφληση. Καταφέραμε να εξασφαλίσουμε τα 5 δισεκατομμύρια, όπως είπατε, δεν θα πήγαιναν στους εθνικούς προϋπολογισμούς. Και πάνω από 4 δισεκατομμύρια ευρώ τα εξασφαλίσαμε για το 2015 και θα πρέπει να τα ξανά ε, χρησιμοποιήσουμε, να τα βάλουμε στον προϋπολογισμό, να αποφύγουμε την κατάρρευση του προϋπολογισμού με, την, ε, με τα ποσά αυτά τα 4,8 δισεκατομμύρια. Η Κομισιόν μπορεί να εξασφαλίσει, να σταθεροποιήσει τα ποσά προς εκταμείευση, το χρέος της λοιπόν, και να παραμείνουμε στα πλαίσια των δημοσιονομικών προοπτικών. Είναι λοιπόν μια καλή λύση. <clears throat> Καταφέραμε να έχουμε πρόσθετους πόρους για να μειώσουμε το χρέος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αν φυσικά είχαμε πάρει την αντίθετη κατεύθυνση, είχαμε καταψηφίσει αυτή τη συμφωνία, αυτό θα σήμαινε ότι τα κρατημέλη ούτε θα μας έδιναν αυτά τα χρήματα και θα έπαιρναν και τα πρόσημα τα 5 δισεκατομμύρια πάλι πίσω. Θυμάστε ότι το Συμβούλιο εξάλλου ήθελε να περικόψει 2,1 δισεκατομμύρια από τη θέση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και καταλήξαμε μονάχα σε 923 εκατομμύρια ευρώ περικοπών. Επίσης, ενισχύουμε και ορισμένε γραμμές του προπολογισμού που είναι πάρα πολύ σημαντικές για την ανάπτυξη και την απασχόληση και ιδίως στην κατηγορία 1α με προγράμματα όπως το COSME, το Horizon 2020 και την κατηγορία 4 η οποία περιλαμβάνει την ανθρωπιστική βοήθεια. <clears throat> και στην αρχή των διαπραγματεύσεων όπως είχε τονιστεί και από πολλούς. Αυτό το οποίο ήταν πάρα πολύ σημαντικό ήταν το να εξασφαλίσουμε ένα σχέδιο για τη μείωση του χρέους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή των εκκρεμουσών πληρωμών. Είναι απαράδεκτο η Ευρωπαϊκή Ένωση να μην τηρεί τα υπεσχημένα και να έχει ένα τόσο ψηλό επίπεδο πληρωμών οι οποίοι δεν εξοφλούνται. Εδώ το κοινοβούλιο λοιπόν έπρεπε να μαζέψει τα μπάζα, αν μπορώ να το πω έτσι, και έπρεπε να επιβάλλει στην Κομισιόν και το Συμβούλιο να κάνουν τα απαραίτητα. Εδώ πρόκειται απλώς για μια εφαρμογή των συνδικών και εξόφλησης των χρεωστουμένων, ανάληψης πλήρους των υποχρεώσεών μας. Αυτή λοιπόν η συμφωνία είναι πάρα πολύ σημαντική και εξασφαλίζει ότι θα υπάρξει ένα σχέδιο για τις πληρωμές που οφείλονται χωρίς να τεθεί ένα αμφιβόλο το σύνολο των δημοσιονομικών προοπτικών και των υποχρεώσεων που έχουμε για συγκεκριμένα προγράμματα. Θέλω λοιπόν να συγχαρώ όλους αυτούς που συνέβαλαν σε αυτό το αποτέλεσμα. Έχουμε καταλήξει σε μια καλή συμφωνία <clears throat> η οποία εξασφαλίζει την, την ε, αξιοπιστία της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιτρέπει το 2015 ο προϋπολογισμός ένας προϋπολογισμός υπέρ της ανάπτυξης και της απασχόλησης και εξασφαλίζει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση κινείται προς την κατεύθυνση ενός φορέα ο οποίος πρέπει να αναλαμβάνει τις υποχρεώσεις τους μέσα στα δημοσιονομικά πλαίσια. Γι' αυτό και πάλι συγχαρητήρια για όλους και όπως είπα προηγουμένως το να καταψηφίσουμε αυτήν την συμφωνία θα σήμαινε ότι θα ξαναδώσουμε στους εθνικούς προϋπολογισμούς περισσότερα λεφτά και θα θέσουμε τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό σε μεγάλο κίνδυνο. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ, λέει ο πρόεδρος, ο κύριος Μπέιερ. Ευχαριστώ, πρόεδρε. Εγώ να ξεκινήσω από την άλλη. Τι δεν μας ικανοποιεί. Νομίζω ότι ναι μεν καταλαβαίνω ε, τη χαρά σα για τα 3,5 δισεκατομμύρια που δείχνετε παραπάνω, αλλά παρόλα αυτά δεν φτάνουν στι διαπραγματεύσει. Προσπαθήσαμε να αποτρέψουμε μια κατάσταση όπου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτρέχει του Συμβουλίου γιατί θέλει να αποτρέψει τα 12 μορία και έτσι κάνει πιο εύκολες προτάσεις προς το Συμβούλιο. Εγώ σημείωσα ότι τα 4,7 δισεκατομμύρια τα οποία ξεκίνησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ήταν το ποσό όπου θα μπορούσαν να είναι σίγουροι ότι δεν θα συνεχιζόταν το βουνό των χρεών. Πλέον είμαστε στα 3,5 δισεκατομμύρια. Αυτό τι σημαίνει ότι ενδεχομένω να μην φτάσουν τα χρήματα για να σταθεροποιηθούν τα χρέη, τα οποία ενδεχομένω να αυξηθούν και το θέμα των, της χρηματοδότησης των ειδικών μέσων, ούτε αυτό διευκρινίστηκε. Το 2015 μια φυσική καταστροφή να παρουσιαστεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση που θα πρέπει να κινητοποιήσει το Ταμείο Αλληλεγγύης θα σημαίνει ότι θα υπάρξει πάλι κρίση πληρωμών γιατί είτε θα βρούμε τα χρήματα και θα μείνουν απλήρωτοι λογαριασμοί είτε θα μπούμε στη διαδικασία για τα φρέσκα αυτά χρήματα. Θετικό είναι το εξής, ότι το Συμβούλιο πλέον βρίσκεται στην εξής κατάσταση, όπου κάνει σοβαρές διαπραγματεύσεις για τη μείωση των χρεών Αυτό προποθέτει και αναφορά από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα πρέπει τακτικά να μα ενημερώνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το πώ εξελίσσεται η χρήση. Και αν έχω μία προσωπική επιθυμία προ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εκφράσω, θα ήταν η εξή. Θα ήθελα τα χρέη να τα κατανέμουμε και να τα παρουσιάζουμε αναχώρα. Να έχουμε ένα πίνακα στι διαπραγματεύσει που να ξέρω, αν χρειαστεί, και να μπορώ να λέω στον Υπουργό Οικονομικών μου τι Ισχύει. Γιατί στη Γερμανία, για παράδειγμα, να μπορώ να λέμε και για τη Βρετανία, για παράδειγμα, τι ποσά χρωστώνται και πού. Το θέμα δεν είναι να βρισκόμαστε σε πλανεκτική θέση. Το θέμα είναι να μπορούν να πληρωθούν λογαριασμοί και να είναι δικαιολογημένε οι δράσει του Συμβουλίου. Πολιτικά λοιπόν βρισκόμαστε σε μια καλή θετική κατάσταση με σωστά επιχειρήματα, την οποία και πρέπει να αξιοποιήσουμε να βρούμε λύσει. Για το 3,5 δισεκατομμύρια νέα χρήμα είναι πολύ καλή είδηση. Ακόμα και αν ξεκινήσαμε διαφορετικά. Έχει απόλυτα δίκιο ο συνάδελφος. Εμείς είχαμε υποστηρίξει την αξίωση των 4,7 δισεκατομμυρίων. 3,5 δισεκατομμύρια έδωσε το Συμβούλιο και με τους Γερμανούς δημοσιογράφους χθε είχα την τιμή να δούμε πόσο είχαμε τσακωθεί και για ποια ποσά είχαμε τσακωθεί και το 2014. 700 εκατομμύρια μας είχε λοιπόν ε, για 700 εκατομμύρια έχει γίνει ο καυγά πέρσι. Τώρα το Συμβούλιο μας δίνει 3,5 δισεκατομμύρια. Αυτό φυσικά είναι ένα σημαντικό επιχείρημα. Τώρα το περιθώριο για τα πρόβλεπτα έξοδα και αυτό θα πρέπει να κινητοποιηθεί. Γιατί ξεκινάει η κατάσταση να γίνεται ανεξέλεγκτη. Στην ψυχολογία υπάρχουν διάφορα επίπεδα θεραπεία. Ξεκινάμε με το πρόβλημα, μετά υπάρχει αντίσταση. Ε, εμείς έχουμε περάσει πέρα από το στάδιο. Πλέον έχουμε μπει στη φάση της θεραπείας. Σταματάει πλέον η αντίσταση και μπορούμε να ξεκινήσουμε να επιλύουμε το πραγματικό πρόβλημα. Και νομίζω ότι στα τέλη του χρόνου είναι καλή είδηση. Θα ήταν λίγο πιο απλά τα πράγματα όμως για να μπορέσουμε να κάνουμε και εθνική πολιτική. Για το θέμα των πληρωμών. Είναι πάνω από 3,5 δις. Από τα 7 που είναι η διαφορά ανάμεσα σε αυτό το οποίο ζητούσαμε καταρχάς και σε αυτά τα οποία πρότεινε το Συμβούλιο για το 2014 και 2015. Η διαφορά όπως είπα ήταν 7 δις και αυτό το οποίο κερδίσαμε είναι επιπλέον φρέσκο χρήμα κάτι παραπάνω από 3,5 δις το 2014 και 1 δις 200 εκατομμύρια το 2015. Αυτό κάνει 4,8 δις σε σχέση με τα 7 που ήταν η αρχική διαφορά. Ο κύριος Τάγκ, ευχαριστώ πρόεδρε. Θα ήθελα... Μου άρεξε η λέξη που άκουσα ότι ήταν γλυκόπικρη η πραγματικότητα. Κάποια πρόοδο σημειώσαμε αξιόλογη τις τελευταίους μήνες. Για πρώτη φορά το είδα αυτό και βλέπω ποια είναι η αντίσταση από πλευράς του Συμβουλίου που δεν αποδέχεται τη χρήση του περιθωρίου για τα προβλεπτά έξοδα, αρνείται το πρόβλημα των πληρωμών. Νομίζω ότι έχουμε διανύσει μεγάλη απόσταση. Έχουμε θέσει το πρόβλημα επιτάπητος και το έχουν αποδεχτεί οι χώρες. Έχουν αποδεχτεί ότι υπάρχει πρόβλημα και ότι πρέπει να πληρώσουν. Παρόλα αυτά δεν έχει ολοκληρωθεί ο αγώνας αυτός. Ε, θα συνεχιστεί. Και αυτό είναι το πιο πικρό σκέλος, αν θέλετε, της πραγματικότητας. το τελικό αποτέλεσμα λοιπόν αναβάλλεται, θα συνεχιστεί ο αγώνας. Συγγνώμη, ζητάει ο πρόεδρος. Συνεχίστε κύριε Τάγκ. Χαίρομαι λοιπόν ε, σε ό,τι αφορά το σχέδιο πληρωμών. Είναι κρίσιμη σημασία για να συνεχίσουμε να ασκούμε πίεση και προκειμένου να καταστεί το πρόβλημα των πληρωμών πιο διαχειρίσιμο. Είναι όντως ε, γκρίζα η ζώνη για το κατά πόσο θα έπρεπε να είναι 4,8 δισεκατομμύρια. Πόσο είναι ακριβώς, δεν ξέρουμε ακριβώς τι γίνεται. Είναι λοιπόν καιρός να βγούμε από την θέα αυτή η ζώνη. Και επίσης μας άρεσε και η ιδέα του Γιέντς, του να ξέρουμε τι χρωστάνε συγκεκριμένα οι χώρες, να το ξέρουμε αυτό από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στη δική μου περίπτωση θα ήταν πάρα πολύ χρήσιμο αυτό για το κοινό. Θα πρέπει να είναι πιο προβλέψιμο και πιο διαφανής η κατάσταση. Αυτό είναι σπουδαία σημασία. Να πω και κάτι άλλο στην Επιτροπή αυτή. Γιατί αυτή η διαδικασία δεν έχει να κάνει με το Κοινοβούλιο ούτε με την Επιτροπή μας. Πρόκειται για την ε, συνεισφορά ανα, εισόδημα κατά κεφαλή. Αφενός λοιπόν θέτουμε το πρόβλημα των πληρωμών στην ημερήσια διάταξη. Κάναμε αυτή την κίνηση. Αλλά από την άλλη χάνουμε ως Ευρωπαϊκή Ένωση, τουλάχιστον στην Ολλανδία και για το Ηνωμένο Βασίλειο, γιατί για κάποιους η κατάσταση αυτή είναι απαράδεκτη. Και Ακούμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι οι χώρε θα έπρεπε να το περιμένουν αυτό. Αλλά το γεγονό είναι ότι η κατάσταση είναι τόσο περίπλοκη που πραγματικά οι χώρε ε, βρίσκονται προεκπλήξεω. Και αυτό έχει να κάνει με την ε, πολυπλοκότητα του συστήματο, την ε, διαφάνεια που χρειαζόμαστε. Χρειαζόμαστε διαφάνεια, χρειαζόμαστε προβλεψιμότητα. Βρισκόμαστε σε μια κατάσταση η οποία πραγματικά είναι πολύ δύστη και είναι κρίμα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ετσενίγε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κατανοώ ότι ήταν δύσκολες διαπραγματεύσεις, ιδίως όταν υπάρχει διαπραγμάτευση με ένα τόσο δύσκολο φορέα όπως είναι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Πιστεύω όμως ότι η συμφωνία που επετεύθη είναι η ενδιάμεση λύση ανάμεσα σε δύο ακραίες πλευρές, δύο ακραίες απλό, απόψεις. Μπορούσαμε ίσως να επιτύχουμε περισσότερο, αλλά την απόρριψη δεν θα μπορούσαν να την καταλάβουν οι πολίτες Ευρώπης λέτε, αλλά κρίμα που πρέπει να το πω, στη χώρα μου έχουμε 25% ενεργεία, έχουμε εκατομμύρια ανθρώπων που ζουν με λιγότερο από 300 ευρώ το μήνα. Το χρηματιστήριο στη Γερμανία αυτή τη στιγμή όμως ανεβαίνει συνέχεια. Αν η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μια εμπορική ένωση και τίποτα παραπάνω και το μόνο εργαλείο αναδιανομής πόρων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και της μείωσης των ε, διαφορών που υπάρχουν σε παραγωγικότητα είναι απλώς ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός. Αλλά αυτός ο προϋπολογισμός είναι όλο και πιο μικρός. Το μόνο το οποίο πετυχαίνουμε είναι να αυξάνει οι ανισότητες στην Ευρώπη, το χάσμα μεταξύ των χωρών στην Ευρώπη να είναι μεγαλύτερη σε ό,τι αφορά την ε, προστιθέμενη αξία στην παραγωγή τους αυτό ουσιαστικά είναι έφορο χωράφι για σπορά ιδεών ευρωσκεπτικισμού και βλέπουμε συνέχεια να ανεβαίνει ο ευρωσκεπτικισμός και η αντίθεση προς την Ευρώπη. Πιστεύουμε λοιπόν ότι ξεπεράσαμε τα φαντάσματα του παρελθόντος όπως τα φαντάσματα του φασισμού αλλά κινδυνεύουν να επανέλθουν στο πλαίσιο αυτό που βρισκόμαστε όταν εμείς αντιμετωπίσουμε αυτά τα προβλήματα χωρίς την απαραίτητη ευθύνη. η συγγήτρια μπορούμε να το δούμε το ποτήρι μισοάδιο ή μισογεμάτο, δυστυχώς. Πιστεύω ότι οι πολίτες της Ευρώπης το βλέπουν αυτή τη στιγμή τελείως άδειο το ποτήρι. Ευχαριστώ πολύ. Διευκρινίσω εδώ ότι η Επιτροπή θα συνεδριάσει τη Δευτέρα το βράδυ στο Στρασβούργο στις 7 ε, το απόγευμα για να πάρει αποφάσεις για τον προϋπολογισμό του 2015 και για τις τροπολογίες οι οποίες δεν είχαν ψηφιστεί μέχρι τώρα στον προϋπολογισμό του 2014. Ο κύριος Μάνκα έχει ζητήσει το λόγο. Ε, ε, Σα ευχαριστώ πάρα πολύ Πρόεδρε. Θα ήθελα να συγχαρώ όλη την ομάδα της οποίας και ηγηθήκατε εσείς, Πρόεδρε, αλλά και οι συγητές μας. Ήταν πραγματικά ομαδικό το έργο και το αποτέλεσμα και μπορεί οι απόψεις μας να ήταν διαφορετικές, αλλά σε ό,τι αφορά την εξωτερική διάσταση, το πώς μας αντιλήφθηκε ο κόσμος, επιδείξαμε ένα ενιαίο μέτωπο. Αν δεν είχαμε συμφωνήσει και είχαμε προσωρινά 12 δεν θα είχαμε καταφέρει ούτε το επενδυτικό σχέδιο, ούτε τίποτε άλλο. Θα είχαμε χάσει και όλο το σύστημα θα είχε καταρρεύσει. Μπορεί το σύστημα των προσωρινών των να ήταν καλό για να πληρώσουμε τον, τους λογαριασμούς, δεν θα υπήρχαν νέες επενδύσεις, αλλά θα ήταν πραγματικά αποτυχημένος τρόπος και συμφωνώ με το Γιέντς ότι είναι δύσκολο για μας να σταθεροποιήσουμε το επίπεδο των χρεών. Θα έπρεπε να είναι πιο εύκολο στην αρχή μιας δημοσιονομικής περίοδου, γιατί δεν θα είχαμε τόσο υψηλό επίπεδο εφαρμογής όσο στη μετέπειτα φάση της προγραμματικής περίοδου. Αλλά αν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας ε, καταθέσει ένα χρονοδιάγραμμα για την πληρωμή των χρεών μέχρι το Μάρτιο, θα πρέπει να είμαστε βέβαιοι ότι θα συμπεριληφθεί και ένας πίνακας αναχώρα. Αναχώρα για να ξέρουμε τι χρωστάει κάθε χώρα. Δεν θέλουμε οι χώρε τα κράτη-μέλη, να περιέλθουν σε δύσκολη κατάσταση κάποια από τα νέα κράτη-μέλη, λόγω ακριβώς της χρέωσης αυτής, δεν ε, είναι καθαροί δικαιούχοι πλέον, αλλά καθαροί εισφορείς στον κοινοτικό προϋπολογισμό. Το αποτέλεσμα λοιπόν ήταν το καλύτερο που μπορούσαμε να πετύχουμε, αλλά για το μέλλον θα πρέπει να κάτσουμε και να σκεφτούμε πώς θα δημορφωθεί διαφορετικά η ροή εσόδων για τον κοινοτικό προπολογισμό ανεξάρτητα από την καλή θέληση των κρατών μέλων και από τον εκάστοτε ηγετών τους. Θα πρέπει να καταρτίζουμε ένα προπολογισμό βάσει ιδίων πόρων. Ευχαριστώ η κυρία Βαναάρτ. Τελευταία και μετά θα δώσουμε το λόγο που θα σας διαβέωσει για την σταθεροποίηση και την εισφορά των εσόδων. Έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, Πρόεδρε. Η κυρία εισηγήτρια είπε στην αρχή ότι μπορούμε να δούμε το ποτήρι μισογεμάτο ή μισοάδιο. Ζητώ συγγνώμη αγαπητοί συνάδελφοι, από δική μου πλευρά και από πλευρά τη ομάδα μου θα πρέπει να πω ότι το ποτήρι είναι στεγνό και θα πεθάνουμε από δίψα. Αν μου επιτρέπετε να συνεχίσω τη μεταφορά. Φυσικά ξέρω ότι ήταν πολύ σοβαρέ οι διαπραγματεύσει και ότι ήταν πάρα πολύ ε, μεγάλε οι προκλήσει που αντιμετωπίσαμε. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι' αυτό. Και θα πρέπει να ομολογήσω ότι είμαι και εγώ καινούρια εδώ στο Κοινοβούλιο. Πρώτε διαπραγματεύσει λοιπόν είναι αυτέ που είδαμε. Αλλά το αποτέλεσμα να σας πω ότι ήταν πάρα πολύ απογοητευτικό. Γι' αυτό λοιπόν από δική μας πλευρά θα ήθελα να τονίσω ότι ο προπολογισμό του 2015 δεν μα βρίσκει σύμφωνο. δεν θα τον υποστηρίξουμε. Είναι πολύ πιο κάτω από τι ε, προσδοκίε μα, το είπε και ο συναδελφο Γκάιερ. Ε, μπορεί να μην φτάσει καν. Αυτή είναι η δική μα ανάλυση. Η δική μα ανάλυση μάλλον είναι ότι δεν πρόκειται να φτάσει σε καμία περίπτωση. Το γερμανικό αποτέλεσμα, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τι πληρωμές, είναι 5 δισεκατομμύρια κάτω από την ε, θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. ένα δισεκατομμύριο πάνω από τις εκτιμήσεις του Συμβουλίου. Είναι καλός συμβιβασμός τώρα αυτός. Και φυσικά οι επιτυχίες ε, του 2014 μπορεί να θεωρήσει κανείς ότι αποτελούν επιτυχίες. Αλλά αυτό αντισταθμίζεται από τα επόμενα κρατημέλη και η, τα έξοδα των κρατών μελών, η χρέωση των κρατών μελών θα είναι πιο μεγάλα από την αύξηση του προπολογισμού. Αυτό να το λάβουμε υπόψη. Το πιο πικρό ποτήρι για μας είναι το θέμα των ε, πληρωμών που δεν έχουν πληρωθεί. Δεν σταθεροποιήθηκε καν το θέμα αυτό των απλήρωτων ε, λογαριασμών. Έχει επιδεινωθεί περαιτέρω η κατάσταση. Και όπως συχνά το συζητήσαμε στην Επιτροπή μας, αυτό διακυβεύει και υπονομεύει την εμπιστοσύνη σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πόσο μάλλον σε ό,τι αφορά τους επιχειρηματίες. Καθόλου κανοποιητική κατάσταση. Να αναφερθώ και σε αυτά που είπε ο πρώην Επιτροπός και πλέον συνάδελφος Λεβαντόφσκι. Να συμφωνήσω γιατί μας προειδοποίησε ότι ο προϋπολογισμός αυτός θα μας οδηγήσει σε απώλεια ενδεχομένως του τριπλού α από τους οργανισμούς πιστοληπτικής ικανότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι τουλάχιστον ανησυχητική η κατάσταση και πολύ απογοητευτική η κατάσταση σε ό,τι αφορά το αποθεματικό του προπολογισμού που για πρώτη φορά δεν χρησιμοποιήθηκε από τον Ευρωπαϊκό, από τον, από την Ευρωπαϊκή, από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε ό,τι αφορά την ομάδα των εμπειρογνωμόνων σε φορολογικά θέματα τα μεγάλα τέσσερα κόμματα εδώ στο Κοινοβούλιο μπορεί να κάτσουν και να συνεχίσουν, για παράδειγμα, τα ίδια άτομα προκάλεσαν τα φορολογικά ζητήματα φορολογική αποφυγή, φοροδιαφυγή και αποφυγής στο Λουξεμβούργο να συνεχίσουν να ε, δουλεύουν ως σύμβουλοι στο Ευρωπαϊκό, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ. Τη Δευτέρα το βράδυ θα έχουμε την ευκαιρία για να συμφωνήσετε, να διαφωνήσετε με τα συμπεράσματα του τριγωνικού διαλόγου. Κάποια καταπραγητικά τώρα λόγια για να σας πείσω ότι το χρέος έχει σταθεροποιηθεί και θα αρχίσει από το 2015 να μειώνεται. Κύριε Καλβίνιο από την Κομισιόν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα τέσσερα σημεία να αναφέρω. Και πράγματι ελπίζω ότι αυτά τα οποία θα σας πω θα μας επιτρέψουν να καταλήξουμε στη συζήτηση αυτή με αισιόδοξο τρόπο. Έρχονται γιορτές άλλωστε. Ξεκινώντας, ε, η λύση στην οποία καταλήξαμε νομίζω ότι είναι μια πολύ ισορροπημένη λύση. Συνειδητοποιούμε πλέον ότι οι υποχρεώσεις θα πρέπει να γίνονται σεβαστές και τα προγράμματα θα πρέπει να εκτελούνται στην ολότητά τους. Θα πρέπει επίσης να συνειδητοποιούμε ότι τα χρήματα δεν τα κόβει κανείς από τα δέντρα, προέρχονται από τους πολίτες, από τις επιχειρήσεις, από τους φόρους και ιδιαίτερα σε δύσκολους καιρούς, γιατί ξέρετε ότι υπάρχουν πολλές χώρες που αντιμετωπίζουν δύσκολες δημοσιονομικές καταστάσεις. Συνεπώς η ισορροπία είναι μια καλή ισορροπία, μια θετική ισορροπία. Να μου επιτρέψετε να προσθέσω ορισμένα επιπλέον στοιχεία σε σχέση με αυτά τα οποία είπαν οι εισηγητές και που περιλαμβάνονται φυσικά στη συμφωνία. Ένα πρώτο στοιχείο που αφορά τις ανησυχίες για τις πληρωμές είναι ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή σχέση πληρωμών και υποχρεώσεων 97% περίπου το 14 και το 15 κάτι το οποίο είναι πολύ ικανοποιητικό, πολύ περισσότερο από το παρελθόν. Οι πληρωμές έχουν διατηρηθεί για το 1α, για το 4, και για τη σύγκληση και τη συνοχή, που είναι οι πολιτικές προτεραιότητες και για σας και για την Ευρώπη τελικά. Αν διαβάσει κανείς τις κατευθυντήριες ε, γραμμές οι οποίες προέρχονται από το Συμβούλιο. Από πλευράς Κοινοβουλίου έχετε παραδεχθεί ένα σημαντικό ποσό για τα προπαρασκευαστικά και πιλωτικά προγράμματα και κάποιες από τις προτάσεις του Κοινοβουλίου έγιναν δεκτές και ε, γύρω από τις εξωτερικές υπηρεσίες και τους άλλους οργανισμούς. Θα ήθελα επίσης να υπογραμμίσω ένα θέμα το οποίο σε κάποια φάση ήταν πολύ σοβαρό πολιτικό πρόβλημα και το οποίο το έχουμε παραμερίσει εν τώρα. Καταφέραμε να αντιμετωπίσουμε τις ανάγκες συνέπειες του ρωσικού εμπάργου στη Γεωργία. Αυτό είναι σημαντικό για όλα τα όργανα και κυρίως φυσικά για τους ίδιους τους γεωργούς. Και νομίζω ότι οι προϋπολογισμοί αυτοί θα επιτρέψουν την σταθεροποίηση και μείωση των απλήρωτων λογαριασμών, του άχθους του παρελθόντος. Αν εξετάσουμε λοιπόν τα στοιχεία των εισηγητών και τα επιπλέον στοιχεία που ακούσαμε, η ισορροπία πρέπει να είναι ικανοποιητική. Μία επιπλέον σκέψη είναι ε, η εξής. Να μου επιτρέψετε να πω ότι σε μία περίοδο προϋπολογισμού, σε έναν ετήσιο προϋπολογισμό, όλα τα προβλήματα της Ευρώπης δεν θα μπορέσουμε να τα λύσουμε. Θα έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας τα επόμενα χρόνια, θα έχουμε πάρα πολλή πίεση για το 2015, ήδη από τις αρχές του 2015 θα πρέπει να φτιάξουμε ένα πρόγραμμα, ένα σχέδιο πλήρωμων, θα υπάρξουν πολλές συζητήσεις που θα ακολουθήσουν το 2015 με μεγάλη ένταση. Θα χρειαστεί να αναπρογραμματίσουμε τα τα ταμεία στα οποία δεν υπήρξε συμφωνία μετά το τέλος του 2014. Θα πρέπει επίσης να δούμε τι δημοσιονομικές συνέπειες θα πρέπει να υπάρξουν ή θα υπάρξουν από το πρόγραμμα επενδύσεων ε, Juncker και τι νομική βάση θα χρησιμοποιηθεί Όλα αυτά θα επανέλθουν και όλα αυτά θα συζητηθούν ξανά και ξανά. Κάτι το οποίο προκαλεί, καταλαβαίνω, μια κάποια δυστημία. Μια τελευταία σκέψη εδώ. Θεωρούμε ότι δεν νίκησε το ένα όργανο και έχασε το άλλο. Και τελικά αυτό είναι και λίγο άσχετο θα ήθελα να πω. Αυτό το οποίο επιδιώξαμε είναι να καταλήξουμε σε μια συμφωνία θετική για τις επιχειρήσεις, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τους πολίτες. Αυτό σημαίνει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να τιμήσει τις προτεραιότητες της, τις υποσχέσεις της. Οι ανησυχίες μας δεν ήταν τα προσωρινά 12 τιμωρία. Η ανησυχία μας ήταν οι πολίτες να δουν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να βρει λύσεις στα προβλήματα. Δημιουργούμε ένα σταθερό δημοσιονομικό πλαίσιο. Δεν είναι το καλύτερο δυνατόν, αλλά θα αυξήσει τη σταθερότητα, θα αυξήσει την αίσθηση γενικά εμπιστοσύνη στην Ευρώπη. Αυτό δεν θα μπορούσαμε να το κάνουμε χωρίς τη δική σας αποφασιστικότητα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί παίξατε ένα εξαιρετικό ρόλο και θα συνεχίσετε να παίζετε ένα εξαιρετικό ρόλο τα επόμενα χρόνια έτσι ώστε να έχουμε ένα καλό προϋπολογισμό στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Merci. Σας ευχαριστώ λέει ο Πρόεδρος. Ο καθένας θα έχει τη δική του άποψη για τα γεγονότα αυτά. Ε, θα ήταν ίσως ε, πάρα πολύ υπερβολικό να θεωρήσουμε ότι έχουμε λύσει όλα τα προβλήματα. Έχει ξεκινήσει η διαδικασία, όλα εξαρτώνται από την αποφασιστικότητά μας, από τη δέσμευσή μας να μπορέσουμε να λύσουμε σταδιακά το πρόβλημα αυτό. Αυτό το οποίο ζήσαμε θα πρέπει να μας οδηγήσει σε κάποιο προβληματισμό. Έχουμε όλα τα στοιχεία για να προχωρήσουμε σε ένα σεμινάριο προϋπολογιστικού αναστοχασμού προς το τέλος Ιανουαρίου, ίσως με τον τρόπο αυτό φτάνουμε και στο τέλος ενός κύκλου του προϋπολογισμού και είναι πολύ ενδιαφέρον να κατανοήσουμε ότι έχουμε περάσει όλο μας το χρόνο στη διαπραγμάτευση για τις πιστώσεις πληρωμών και δεν έχουμε αρκετή σκέψη για το μέλλον. Και Φυσικά εμείς έχουμε εκλεγεί πρόσφατα. Βρισκόμαστε πολύ κοντά στην ενδιάμεση αναθεώρηση των δημοσιονομικών προοπτικών 2014-2020. Αυτό είναι το μεγάλο ραντεβού. Θα πρέπει να προετοιμαστούμε καλύτερα για τα θέματα αυτά και για τις πληστώσεις πληρωμών θα έχουμε την ευκαιρία να ανταλλάξουμε απόψεις και στο μέλλον. Είχαμε την ένδειξη των πληρωμών που οφείλονται σε κάθε χώρα, το είχαμε δει στο παρελθόν και φαντάζομαι ότι και για το τέλος του 2014 μας δώσει η Κομισιόν ένα νέο έγγραφο. Πρέπει να σκεφτούμε και για την αποτελεσματικότητα των δημοσίων δαπανών, γιατί όλοι καλούμαστε να τις συμπιέσουμε. Πρέπει να δούμε και ποιος είναι ο πραγματικός αντίκτυπος επιτοπίως. Είναι πολύ εύκολο να πούμε από τις Φρυξέλλες ότι θα πληρώσουμε τους, ε, αυτούς που εκτελούν τα προγράμματα αργότερα, αλλά αυτοί το αντιμετωπίζουν πολύ πιο βαριά και αυτό αυξάνει τον, αυτοσκεπ... τον ευρωσκεπτικισμό. Το θέμα δεν είναι επίσης να δούμε αν κέρδισε το Κοινοβούλιο, το Συμβουλίο ή η Κομισιόν. Αυτό το οποίο είναι απαραίτητο είναι να κερδίσει η Ευρώπη <clears throat> και οι Ευρωπαίοι. Τούτων λεχθέντων, νομίζω ότι μπορούμε να κλείσουμε τη συζήτηση αυτή και όπως σας είπα θα πάω στη συνέρευση των Προέδρων. Καλό τον κύριο Γκάιερ να αναλάβει την Προεδρία της Επιτροπής μας γιατί θα πρέπει να ακούσουμε τον εισηγητή μας τον κύριο Λεβαντόφσκι και τον κύριο Ντεπρέ για την επιταχυμένη διαδικασία. Η διαδικασία αυτή τουλάχιστον θα πρέπει να είναι ένα στοιχείο το οποίο θα έχει το ρόλο νομολογίας. Όπως είπαμε στις, ε, στη συζήτηση για τις δημόσιες αγορές, χρειαστήκαμε τρία χρόνια για να αλλάξει η ρύθμιση. Εδώ έχουμε πετύχει όμως πολύ γρήγορα μια αλλαγή των κανόνων και αυτό οφείλεται στην πολιτική μας θέληση. Σας εύχομαι λοιπόν κάθε επιτυχία στη συνέχεια των συζητήσεων και θα τα πούμε τη Δευτέρα στις 7 το βράδυ στο Στρασβούργο. Κύριε Γκάιερη, παίρνετε την έδα μου. Οπότε, αγαπητοί συνάδελφοι, με κάποια καθυστέρηση περνάμε στο επόμενο σημείο της σημερινής διάταξης. τροποποιητικός κανονισμός, ο οποίος τροποποιεί το κανονισμό σε σχέση με τους ίδιους πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο κύριος Ντεπρέ και ο κύριος Λεβεντόφσκι είναι οι Κύριε Λεβαντόφσκι, θέλω να σας ευχαριστήσω. Συγχαρητήρια σε όλους αυτούς που έλαβαν μέρος στη συνδιαλλαγή. Ήταν πολύ δύσκολο αυτό το έργο. Είναι όμως το θέμα του τι μπορεί κανείς να επιτύχει, τι είναι εφικτό και όχι απλώς τι είναι επιθυμητό. Τώρα αντιμετωπίσουμε την δεύτερη επιστολή του Συμβουλίου για να δώσουμε την ε, ε, να δώσουμε την έγκρισή μας στην καθυστέρηση της καταβολής των ε, οφειλωμένων ποσών στον προπολογισμό από ορισμένα κράτη. Την πρώτη φορά υπήρξε μια άρνηση. Τώρα έχουμε ένα πακέτο για το 2014-2015. Μπορούμε λοιπόν να μομιμοποιήσουμε την αναβολή των πληρωμών αυτών με τρόπο αναδρομικό. Και είναι έτοιμη λοιπόν η πρότασή μας να ψηφιστεί. Έχουμε δύο τροπολογίες στο ψήφισμα <clears throat> για το νομικού χαρακτήρα κείμενο και εμείς ε, τονίσουμε την ανάγκη να γίνουν διάφανα τα στοιχεία που έχουν να κάνουν με την αναβολή. Είχαν κατατεθεί 17 τροπολογίες σχετικά, τρεις από αυτές έχουν αποσυρθεί έκτοτε, έξι από τους εισηγητές. Είναι μια κατεπίγουσα διαδικασία, θα πρέπει να ψηφίσουμε την επόμενη εβδομάδα στο, στην Ολομέλεια. Εγώ δεν θέτω το θέμα του αν ήταν πράγματι κατεπίγουσα ή όχι η διαδικασία αυτή. Αυτό που είναι απαραίτητο είναι να νομιμοποιήσουμε την επόμενη εβδομάδα αυτό το οποίο ζητήθηκε για τα κατημέρια της αναβολή της καταβολής πληρωμών. Δεν Κύριε Ντεπέ, ευχαριστώ πρόεδρε. Δεν θα προσθέσω τίποτα στα λεγόμενα του κυρίου Λεβαντόσκη. Μόνο ότι στις συμφωνίες τις οποίες καταλήξαμε προβλέπεται να ψηφίσουμε την πρόταση αυτή, όσοι την στηρίξουν εν πάση περιπτώσει, γιατί είναι τμήμα του πακέτου. Η, το περιθώριο κίνησης το οποίο έχουμε είναι περιορισμένο πλέον εδώ, εφόσον θέλουμε να παραμείνουμε στα πλαίσια των προηγούμενων αποφάσεων. Σα ευχαριστώ πολύ. Δεν ξέρω αν ζητάει κανείς άλλο το λόγο για το θέμα αυτό. Δεν βλέπω κανένα να ζητάει το λόγο και θα κάνουμε την ε, ψηφοφορία λοιπόν κατευθείαν και θα αποφασίσει το Δεκέμβριο η Ολομέλεια. Να περάσουμε στην ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το σχέδιο του επενδυτικού της Ευρώπης. Αυτό ασφαλώς και θα έχει επιπτώσεις για τον προϋπολογισμό και περνάμε λοιπόν σε μια ανταλλαγή απόψεων. Έχουμε λοιπόν μια παρέμβαση καταρχάς από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η κυρία Γενική Διευθύντρια έχει το λόγο. I'm not sure of the... Δεν είμαι βέβαιη αν κατάλαβα καλά. Ναι, το επενδυτικό πρόγραμμα θέλετε να σας παρουσιάσω. Ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ λοιπόν που μας δίνετε την ευκαιρία να κάνουμε μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων και πάλι πιστεύω ότι πρόκειται για ένα θέμα το οποίο θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε σε διάφορες άλλες περιστάσεις του χρόνου, αλλά όντως αποτελεί μία από τις νέες προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και γι' αυτό λοιπόν καλό θα είναι το Κοινοβούλιο να αρχίσει να κάνει σκέψεις και να συμμετέχει στις συζητήσεις και στις σκέψεις αυτές και η Επιτροπή σας. Από πλευράς ε, δικής μας έχουμε ανταποκριθεί σε μία από τις πιο μεγάλες δεσμεύσεις που ε, ανέλαβε ο κύριος Γιούγκερ και εδώ στο Κοινοβούλιο ένα πρόγραμμα επενδυτικό για να υπάρξουν πάνω από 300 εκατομμύρια, εκατομμύρια επενδύσεις επιπλέον στην Ευρώπη. Τα τελευταία χρόνια είδαμε πολύ αρνητικές τάσεις, όπου οι επενδύσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν πέσει σημαντικά από το maximum που είχαν φτάσει το 2007, πτώση πάνω από 15% και αυτό το έχουν εντοπίσει και οι πιο πολλοί αναλυτές ως ένα από τα βασικά εμπόδια για την ανάπτυξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το πρόγραμμα ε, περιέχει και ένα δημοσιονομικό στοιχείο, θα επανέλθω και στο θέμα αυτό, αλλά υπάρχουν και άλλα δύο στοιχεία. Εντοπισμό ροών επενδύσεων και προγραμμάτων που μπορεί να έχουν μεγάλη σημασία για την ανάπτυξη και τις θέσεις εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στις υποδομές και ως ενίσχυση στις ε, μικρομεσαίες. Και κατά δεύτερον, καλύτερο ρυθμιστικό πλαίσιο κατάργηση των εμποδίων στις επενδύσεις. Σημαντικά είναι και τα χρήματα, αλλά σε μερικές περιπτώσεις από πλευράς ε, νομοθετικής ε, μας δυσκολεύουν πολύ κάποια εμπόδια όπως η υπερβολική γραφειοκρατία. Η, Επιτροπή προφανώς η δική σας θα ενδιαφέρεται ιδίως για τα δημοσιονομικά στοιχεία. Ευρωπαϊκό Ταμείο λοιπόν για στρατηγικές επενδύσεις, βασικό στοιχείο, το οποίο θα δημιουργηθεί για να υπάρξει υποστήριξη σε ό,τι αφορά το ρίσκο μακροπρόθεσμων επενδύσεων και για τη μείωση του κινδύνου για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Η ιδέα είναι να υποστηριχθούν προγράμματα υποδομών σε βριζονικότητα, μεταφορές, αλλά το τονίζω αυτό γιατί πιο πολλοί ε, εστιάζονται σε θέματα υποδομών, αλλά εμάς μας ενδιαφέρουν και οι υποδομές οι κοινωνικές, όπως η εκπαίδευση, η ενέργεια, η ενεργειακή αποδοτικότητα. Και ο πρόεδρος Ιούνκερ δίνει ιδιαίτερη σημασία. Δεν θα υπάρχουν θεματικές ή γεωγραφικές προ, ε, κατανομές, πρώτερες κατανομές. Δεν μιλάμε για το άθροισμα 28 επενδυτικών σχεδίων. 240 δισεκατομμύρια λοιπόν θα δαπανηθούν σε αυτές τις υποδομές και 75 δισεκατομμύρια θα κινητοποιηθούν σε ό,τι αφορά τις επενδύσεις σε μικρομεσαίες. Η διαδικασία αυτή θα είναι με ανοιχτό ορίζοντα για να ολοκληρωθούν τα έργα αυτά και το Ταμείο θα εδρεθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Επενδυτική Τράπεζα. Ξέρω ότι είναι εδώ πέρα ένα συνάδελφο από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων που μπορεί να πάρει το λόγο αν υπάρχουν συγκεκριμένε ερωτήσει προ αυτόν και θα υπάρξει μια ανεξάρτητη Επιτροπή Επενδύσεων που θα εξετάσει την βιωσιμότητα και την προστιθέμενη αξία των μεμονωμένων προγραμμάτων προς επένδυση προσχηματοδότηση. Από πλευράς ευρωπαϊκού προϋπολογισμού θα υπάρξει εγγύηση 16 δισεκατομμυρίων ευρώ με δέσμευση 5 δισεκατομμυρίων από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, 21 δισεκατομμύρια λοιπόν συνολικά που θα επιτρέψει στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων να κινητοποιήσει 60 δισεκατομμύρια στις ε, αγορές ε, ένα προς 3 λοιπόν ε, ε, το ποσοστό μόχλευσης, ένα ευρώ προς 3 ευρώ και αυτό θα επενδύεται σε προγράμματα με κατά μέσο όρο συμμετοχή 20%. Και εδώ λοιπόν έρχεται ο πολλαπλασιαστικός παράγοντας του πενταπλώ, που οδηγεί σε μόχλευση 15% συνολικά. Το ταμείο αυτό εγγυήσεων είναι αρκετά παρόμοιο με το, με το Ταμείο για τις Εξωτερικές Δράσεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Γνωρίζετε λοιπόν ποια είναι η μορφή της σύνθεσής τους και για να υπάρξει αντιστάθμιση ενδεχόμενων απώλειων προκειμένου να παίρνει και μεγαλύτερο ρίσκο η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και να χρηματοδοτεί πιο επικίνδυνα προγράμματα, αν θέλετε, θα βάλουμε τον όρο για την εγγύηση αυτή μέχρι και 50% πολύ ψηλό ποσοστό που σημαίνει ότι ο ευρωπαϊκός προπολογισμό θα πρέπει να συμβάλλει με 8 δισεκατομμύρια ευρώ. Επειδή τα πιο πολλά προγράμματα είναι μακροπρόθεσμα, δεν θα πρέπει να υπάρχουν απώλειες και υποχρέωση πληρωμών το 2015, τα πρώτα χρόνια δηλαδή των προγραμμάτων. Ξεκινάει λοιπόν η χρηματοδότηση από το 2016 για να φτάσουμε μέχρι το 2020 το όρο των 8 δισεκατομμυρίων. Και θεωρούμε ότι αυτό μπορεί να χρηματοδοτηθεί στα πλαίσια του πολιετού δημοσιονομικού πλαισίου. Και γι' αυτό λοιπόν προτείνουμε να αναπτυχούν διαφορετικά κάποια μέσα που περιλαμβάνονται στην παρούσα φάση στον ορίζοντα 2020 και στην διευκόλυνση για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και να κινητοποιηθούν τα αιτήσια περιθώρια που προβλέπονται στο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. Αυτά είναι τα βασικά λοιπόν στοιχεία του συστήματος. Η πρώτη αντίδραση από πλευρά των κρατών μελών ήταν εξαιρετικά θετική. Συζητήθηκε στο ΕΚΟΦΗΝ, έκαναν κάποια κράτη-μέλη ήδη ανακοίνωση ότι πρόκειται να συμβάλλουν, γιατί η ιδέα είναι να υπάρχει ένα ανοιχτό σύστημα που θα επιτρέπει στα κράτη-μέλη και στις εθνικές τράπεζες επενδύσεων να συμβάλλουν και να επενδύουν. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Ιανουάριο σκοπεύει να καταθέσει νομοθετική πρόταση, ένα κανονισμό που θα δημιουργήσει το Ταμείο, την, ε, το Ταμείο Αγγίσεων και θα αναφέρει ποια θα είναι το σύστημα. Μέσω συναπόφασης, το Κοινοβούλιο λοιπόν θα έχει να παίξει σημαντικό ρόλο στην νομοθετική αυτή πρωτοβουλία και ελπίζουμε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίο θα συμφωνήσει για μια διαδικασία επιταχυμένη, fast track, προκειμένου να έχει πραγματοποιηθεί το ταμείο αυτό μέχρι τον Ιούνιο του επόμενου έτους. Και προφανώς θα υπάρχει και ένα σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού που θα δημιουργήσει τις απαραίτητες γραμμές του προϋπολογισμού, να υπάρχουν και οι απαραίτητες μεταφορές, αν και δεν θα υπάρχουν πιστώσεις πληρωμών στο πλαίσιο αυτό μέχρι το 2015. Νομίζω λοιπόν θα έχουμε τη δυνατότητα να επανέλθουμε με περισσότερες λεπτομέρειες τον Ιανουάριο αλλά αυτή είναι μια γενική περιγραφή των προτάσεων τις οποίες θα κάνουμε. Σας ευχαριστώ κύριε Γενική Διευθύντρια. Εγώ ήλπιζα να μπορούσατε να μας δώσετε λίγο πιο πολλές λεπτομέρειες σε ό,τι αφορά το θέμα της κατανομής του σχεδίου αυτού, σε ό,τι αφορά τον προϋπολογισμό Σε ποιες ε, παραγράφους του κανονισμού για τον προπολογισμό βασίζεστε λοιπόν και βασιστήκατε. Υπάρχει λοιπόν η ελπίδα να λειτουργήσει όλο αυτό το σύστημα, αλλά αναφέρεστε στο 140, στο 149 το άρθρο. Δεν άκουσα ιδιαίτερα συγκεκριμένε ε, πληροφορίες. Το γεγονός ότι έχουμε συναπόφαση θεωρώ ότι είναι αυτονοήτο και αυταπόδεικτο. Αν βασιζόμαστε στο άρθρο 140 θεωρώ ότι εδώ υπάρχει μια αντίφαση με αυτό που μας είπατε ότι δεν χρειάζεται να αλλάξουμε τίποτα στον προπολογισμό. Πιστεύω ότι υπάρχει μεγάλη ανάγκη τροποποίησης. δεν θα διαθέσουμε ευρωπαϊκούς πόρους για εγγύησεις αν δεν έχουμε τουλάχιστον μία ιδέα για το πόσο υψηλός είναι ο κίνδυνος που θα βαρύνει την Ευρωπαϊκή Ένωση. Καταλαβαίνω λοιπόν ότι στη τελική ανάλυση δεν μπορούμε να εγγυηθούμε για κάθε πίστοση, μόνο για όσες υπάρχει υψηλός κίνδυνος, αλλά το πώς φτάνετε από τα 8 δισεκατομμύρια στα 16 δισεκατομμύρια αυτό το κόλπο θα πρέπει να το εξηγήσουμε σε ό,τι αφορά το το πολλαπλασιαστικό χαρακτήρα, τον διπλό. Αυτά λοιπόν τα ερωτήματα τα οποία είχα και εγώ εξ αρχής. Ζήτησαν το λόγο κάποιοι συνάδελφοι. Να τους δώσω λοιπόν το λόγο. Ο συνάδελφος Λεβαντόφσκι πρώτος. Ε, ευχαριστώ. Κανένας δεν αμφισβητεί το πρόβλημα με τις επενδύσεις στην Ευρώπη αλλά θα πρέπει να δούμε τι συνέβαινε με το 2007. Θυμάστε ότι τότε η Ευρώπη ήταν σε υπερδιέγευση θα έλεγα και υπήρχαν και πληθωριστικοί κίνδυνοι και αυτό οδήγησε σε κάποια στιγμή σε μια κρίση. Θα έχουμε πολλές ευκαιρίες να τα συζητήσουμε στο μέλλον αυτά τα θέματα. Καταρχάς, η χρηματοδοτική αρχιτεκτονική με καταλήτη τον προϋπολογισμό πως από 8 δις ή από 21 δις θα φτάσουμε στα 315. Και η επιλογή των προγραμμάτων επίσης θα πρέπει να είναι ε, τέτοια έτσι ώστε να υπάρξουν κέρδη από τα προγράμματα αυτά. Κάτι το οποίο δεν είναι δεδομένο, σαν παράδειγμα αν επενδύσουμε σε κτηριακές σχολικές εγκαταστάσεις, δεν ξέρω σε ποιο βαθμό κάτι τέτοιο μπορεί να είναι ιδιαίτερα ελκυστικό και για μας και για τον ιδιωτικό τομέα. Έρχομαι στην εμπλοκή του προϋπολογισμού. Δεν είναι κάτι το καινούργιο το να λειτουργήσει σαν καταλήτης ο προϋπολογισμός και να λειτουργήσει η μόχλευση από εκεί και πέρα. Αυτό δεν ξέρω αν μπορεί να γίνει τώρα κάτω από το πλαίσιο των ανώτατων ορίων με τους ιδίους πόρους. Έχει γίνει στο παρελθόν βέβαια για τη βοήθεια για χώρες εκτός Ευρώπης και για τον μηχανισμό σταθεροποίησης για την Ιρλανδία και την Πορτογαλία. Να δούμε λοιπόν τι μπορούμε να κάνουμε, πώς μπορούμε να ξεπεράσουμε το αντότατο όριο, αλλά να μείνουμε πάντα στους ιδίους πόρους. Αυτά είναι βέβαια θέματα που πρέπει να διευκρινίσει ο Γιούνκερ και ο Κατάινεν, γιατί μιλάμε για φρέσκο χρήμα στη συγκεκριμένη περίπτωση και δεν ξέρω σε ποιο βαθμό μπορούμε να το βρούμε στην παρούσα φάση. Ε, ο προϋπολογισμός ήδη από το 2007 έχει λειτουργήσει σαν καταλήτης για τα διάφορα χρηματοδοτικά μέσα που έχουμε χρησιμοποιήσει και νομίζω ότι ο προϋπολογισμός, το σχέδιο του προϋπολογισμού για το 2015 ε, μπορεί να είναι χρήσιμος, μπορεί να δούμε τι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το 2015 και πώς αυτά τα ποσά τα οποία προβλέπουμε σε ορισμένες θέσεις του προϋπολογισμού για το 2015 να τα ονοματίσουμε εκ νέου με διαφορετικό τίτλο και να τα χρησιμοποιήσουμε για αυτό το οποίο είπατε. Θα είναι δύσκολο να βρούμε επίσης επιπλέον πόρους και ιδιαίτερα με το Horizon 2020 είναι και το πώς θα καταναλώσουμε τις πιστώσεις για τα υπάρχοντα προγράμματα και πώς ταυτόχρονα θα μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε τα χρήματα αυτά σαν εγγύηση. Ε, το θέμα των εγγυήσεων. Ξέρει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι υπάρχουν κάποια όρια στα πλαίσια της χρήσης ε, για τις πιστώσεις του Connecting Europe. Πάνω από τρία δις δεν υπάρχουν νομίζω δυνατότητες. Και αυτό το οποίο ε, εκπλήσει εδώ είναι η εκμετάλλευση των ορίων. Υπάρχει μια συμφωνία για τις δημοσιονομικές προοπτικές η οποία είναι δεδομένη και τώρα αυτά τα όρια υποτίθεται θα μεταφέρονται και θα χρησιμοποιηθούν και για την απασχόληση των νέων. Οπότε πώς θα τα καταστήσουμε διαθέσιμα σαν εγγύηση για το πακέτο επενδύσεων. Το βασικό πρόβλημα για τον προϋπολογισμό ο οποίος θα είναι καταλήτης και εγγυητής είναι το που θα βρεθούν κάποιες πιστώσεις οι οποίες και θα χρησιμοποιηθούν για το 15, 16 και 17 και ταυτόχρονα θα χρησιμεύσουν σαν εγγυήσεις. Κοιτάξτε, εγώ εύχομαι ότι καλύτερο στην Επιτροπή για το πρόγραμμά της. Ε, δυστυχώς όμως υπάρχουν ακόμα πάρα πολλές ερωτήσεις, ιδιαίτερα σχετικά με τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. Ο Ράιμερμπεργκ, ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα πρέπει και εγώ να φύγω, οπότε θα κάνω μονάχα σύντομες παρατηρήσεις. Ξεκινώ από το ερώτημα που έθεσε ο Πρόεδρος, το πώς θα αντιμετωπιστούν τα προβλήματα με, το, με τις δημοσιονομικές προοπτικές. Μας είπε η εκπρόσωπος της Κομισιόν ότι ένα μεγάλο μέρος αυτών έχει να κάνει με τη διαδικασία συναπόφασης. Εγώ όμως θα ήθελα να σας προειδοποιήσω. Πολλές φορές έχουμε ζήσει αυτή την κατάσταση στην Επιτροπή Προϋπολογισμών για διάφορες πολύπλοκες διαδικασίες προγράμματα πλαισίου όπου η Κομισιόν και αυτά έγιναν πριν από μερικά χρόνια. Δυστυχώ ο μιλητή μιλάει πολύ μακριά από το μικρόφωνο. Η Κομισιόν δεν έλαβε υπόψη την θέση του Κοινοβουλίου και έδειξε μια ιδιαίτερη εφευρετικότητα σε ό,τι αφορά την ερμηνεία των νομικών διατάξεων για τον προπολογισμό. Το λέω αυτό με ειλικρίνεια, αλλά περιλαμβάνει και μια προειδοποίηση για όλους. Καλό είναι να έχουμε καινοτόμα χρηματοδοτικά μέσα, να δούμε τι είναι εφικτό, τι μπορούμε να επιτύχουμε και να το δούμε θετικά το θέμα αυτό, αλλά πρέπει να είμαστε και ρεαλιστές συγχρόνως. Όταν η Κομισιόν όμως στο τέλος της ε, ε, ανακοίνωσής της λέει ότι αυτό δεν θα έχει καθόλου επιπτώσεις για τις δημοσιονομικές προοπτικές και αν χρειαστεί μπορούμε να κάνουμε μια μεταρρύθμιση κτλ. στις δημοσιονομικές προοπτικές. Αυτή δεν νομίζω εγώ ότι είναι η καλύτερη διατύπωση, αλλά δεν μπορεί να παραβιάσει τα δικαιώματα του Κοινοβουλίου Κομισιόν. Δεν μπορεί λοιπόν να υπάρξει μια τέτοια αντιμετώπιση για τον προπολογισμό η οποία δεν λαμβάνει υπόψη το Κοινοβούλιο. Αναφέρθηκε η μόχλευση η οποία πρέπει να λάβει χώρα για να λειτουργήσει το πακέτο αυτό. Έχουμε ένα πολύ πολύ ζήτημα που από τη μία πλευρά βασίζεται στην ε, δημόσια ε, ε, στις δημόσιες επενδύσεις. Και εμείς αυτή τη στιγμή όμως δεν έχουμε κάτι συγκεκριμένο το οποίο μπορούμε να βγάλουμε από τις ε, συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Νομίζω ότι υπάρχουν όμως πολλά σχέδια που έχουν αναφερθεί, ιδίως στον τομέα των μεταφορών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το ερώτημα λοιπόν δεν είναι <clears throat> αν υπάρχουν χρήματα, το θέμα είναι αν υπάρχουν πραγματικά σχέδια που να μπορούμε να τα υλοποιήσουμε σε ευρωπαϊκό ή σε εθνικό ή ακόμα και σε περιφερειακό επίπεδο. Αυτό πρέπει να κοιτάξουμε λοιπόν προσεκτικά. για να αντιμετωπίσουμε τις ε, προκλήσεις που αναφέρθηκαν στο ρυθμιστικό πλαίσιο και να δούμε κατά πόσο μπορούμε πράγματι να προχωρήσουμε σε ένα τέτοιο φιλόδοξο πρόγραμμα επενδύσεων. Γι' αυτό είναι σημαντικό για μας ως Επιτροπή Προϋπολογισμών να είμαστε δραστήριοι, να είμαστε πραγματιστικοί, αλλά να είμαστε και αποφασιστικοί σε σχέση με τη συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θα πρέπει εμείς να εξασφαλίσουμε ότι αυτά τα προγράμματα θα τύχουν τις σωστές επεξεργασίες και θα περατωθούν εγκαίρως. Όλα αυτά ναι, αλλά όχι με το τίμημα του να χάσουμε την συμμετοχή του Κοινοβουλίου και της Επιτροπής Προπολογισμού που είναι υποχρεωμένοι να συμμετάσχουν στην αντιμετώπιση αυτών των προγραμμάτων. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, σιγά σιγά μαζεύουμε πληροφορίες για την ιδέα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το πώς θα λειτουργήσει αυτό το πρόγραμμα UKER, το πρόγραμμα των επενδύσεων και, και μετά ακόμα και από την παρουσίαση που έγινε κάποιες αμφιβολίες ίσως να απομακρύνθηκαν υπάρχουν και άλλα θέματα όμως τα οποία δεν είναι πολύ ξεκάθαρα και αν χρειαστεί θα κάνω συγκεκριμένες ερωτήσεις ε, στην Επιτροπή. Τώρα για τον προϋπολογισμό. 16 είναι αυτά τα εκατομμύρια, εμείς θα καλύψουμε ε, με 50% και για το 2015 υποτίθεται ότι δεν θα υπάρξουν ε, ε, δημοσιονομικές συνέπειες τουλάχιστον στο επίπεδο των πληρωμών. Δεν θα επηρεαστεί δηλαδή ο προϋπολογισμός τώρα για τις πιστώσεις υποχρεώσεων. Δεν ξέρω πώς θα αντικατοπτρίσετε τις ποσοστώσεις, τις υποχρεώσεις στον προϋπολογισμό του 2015 δεν ξέρω πώς θα χρησιμοποιηθούν κάποια χρήματα με δύο ρόλους. Και αυτό ίσως ε, θα ισχύσει και για τους διορθωτικούς προϋπολογισμούς. Για τη νομική βάση δεν ξέρω αν μπορεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας πει σε τι τομείς εργάζεται, ποια είναι τα θυμία στα οποία ε, θα σταθεί και τι είδους συνεισφορές εθελοντικού τύπου μπορεί να υπάρξουν από τα κράτη-μέλη προς το Ευρωπαϊκό αυτό ταμείο. Δεν ξέρω εφόσον γνωρίζουν ποια θα είναι η στάση των κρατών μελών και τι ποσά είναι αυτά τα οποία θα προσφέρουν. Εφόσον υπάρχει επιθυμία από πλευράς των κρατών μελών ή ορισμένων κρατών μελών να πάρουν μέρος. Επίσης αναφέρθηκε ότι θα μπορούσε να λειτουργήσει κάτι σαν το εξωτερικό ταμείο, ταμείο εγγυήσεων που υπάρχει προηγουμένως από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Όλα αυτά είναι όμως γενικότητες, γενικολογίες αυτή τη στιγμή. Αν θέλουμε να προχωρήσουμε με μεγάλη ταχύτητα θα πρέπει να έχουμε πολύ περισσότερες λεπτομέρειες σε ό,τι αφορά τη συμμετοχή του Ευρωπαϊκού, της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων Αναφέρθηκε επίσης η δημιουργία μιας ανεξάρτητης επιτροπής η οποία θα αξιολογεί τις ε, επενδύσεις, τα σχέδια, αλλά αυτή θα πρέπει να κρίνει τα σχέδια βάσει ποιων κριτηρίων, με ποιο τρόπο θα λαμβάνονται οι αποφάσεις από αυτή την Επιτροπή και ποια θα είναι η σύνθεσή της. Αυτό παραμένει ακόμα ασαφές. Ανεξάρτητη Επιτροπή λοιπόν, αλλά με ποιους. Αυτό είναι λοιπόν το τελευταίο ερώτημα που ήθελα να θέσω προς το παρόν δεν είναι μονάχα το, ο κατάλογος των ερωτήσεων που τελείωσε, αλλά κλείνει και ο κατάλογος των ομιλητών Φερνάντες Μάγκα, Ετσινίκε, Ταράντ και Ντεπρέ. Μπορώ να κλείσω λοιπόν τον μακρό αυτόν κατάλογο. Μπορούμε να θεωρήσουμε ότι έχει κλείσει ο κατάλογος αγορετών. Σας παρακαλώ λοιπόν λαμβάντας υπόψη και το ορολόγιον να περιοριστείτε χρονικά. Ο κύριος Φερνάντης. Θα είμαι σύντομος κύριε Πρόεδρε. Το πρώτο μου ερώτημα είναι με ποιο τρόπο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί να συμμετάσχει περισσότερο στη διαδικασία αυτή ώστε να δοθεί δημοκρατική νομιμοποίηση σε αυτό το σχέδιο επενδύσεων. Αυτό είναι το κεντρικό ερώτημα που με απασχολεί. Το σχέδιο αυτό θα έχει επιπτώσεις στο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Ελέγχθη ότι τα χρήματα αυτά θα χρησιμοποιηθούν, τα 50% των 16 δισεκατομμυρίων θα χρησιμοποιηθούν ως εγγύησης. Αλλά πώς ακριβώς θα χρησιμοποιηθεί αυτή η εγγύηση, τα 8 δισεκατομμύρια, σε ποια χρόνια, σε ποιο κομμάτι των προοπτικών και πόσα χρόνια θα κρατήσει αυτή η εγγύηση εγώ φαντάζομαι ότι τα σχέδια αυτά επενδύσεων μπορεί να έχει μια διάρκεια η οποία μπορεί να ξεπεράσει τις δημοσιονομικές προοπτικές. Θα υπάρχει λοιπόν εγγύηση σε όλη τη ζωή ενός σχεδίου ή θα είναι για δύο ή τρία χρόνια παραδείγματος χάρη. Δεν θα υπάρξουν πληρωμές για τις εγγύησεις αυτές το 2015. Υποθέτω θα ξεκινήσουν από το 2016. Αλλά ήδη στον προϋπολογισμό του 2015 και χωρίς να υπάρχουν αυτές οι πληρωμές υπάρχουν οι αντάβιες αυτού του σχεδίου επενδύσεων του ούτως ελεχθέντων. Το ερώτημα μου είναι ποιες είναι οι προθέσεις για την χρησιμοποίηση στο σχέδιο αυτό επενδύσεων κονδυλίων από τα διαρθρωτικά ταμεία που δίνονται από τα κράτη-μέλη ο κύριος Μάνκα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ λοιπόν κύριε Γιένς. Νομίζω ότι στόχος αυτού του επενδυτικού προγράμματος είναι η χρηματοδότηση επενδύσεων και επενδυτικών προγραμμάτων που παρουσιάζουν κινδύνους και εμείς παρεμβαίνουμε κυρίως για να μειώσουμε τους κινδύνους αυτούς. Πράγματι εμείς χρειαζόμαστε τους ιδιώτες επενδυτές και δεν αρνούμε ότι μπορεί να υπάρξει ρόλος μόχλευσης από πλευράς του προϋπολογισμού. Απαιτούνται επενδύσεις βέβαια κυρίως σε τομείς τους οποίους μπορεί να υπάρξει ε, απόδοση ε, και ταυτόχρονα υπάρχουν και κάποιοι τομείς οι οποίοι δεν είναι και ιδιαίτερα επικίνδυνοι επενδυτικά. Πέρα δηλαδή από τις προτάσεις αυτές θα πρέπει να υπάρξουν και άλλου τύπου επενδυτικές δραστηριότητες. Ένα παράδειγμα, το 40% της ενέργειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση χρησιμοποιείται για την θέρμανση των κτηρίων. Σύμφωνα με την ίδια την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορούμε να μειώσουμε τον όγκο αυτής της ενέργειας στα 3 τέταρτα, κατά 3 τέταρτα συγγνώμη, εφόσον αναλάβουμε δράση σε επίπεδο τεχνολογικό. Να λοιπόν ένας τομέας με μηδενικό κίνδυνο. Είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να αντιμετωπιστεί με την βοήθεια και των ιδιωτικών πιστοτικών ιδρυμάτων. Η τρίτη επιλογή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την απομάκρυνση των εμποδίων ε, στο εμπόριο. Χρειαζόμαστε εδώ κάποια περισσότερη ανάλυση, να δούμε γιατί είδαμε ότι υπήρξε μείωση των επενδύσεων κατά 15% σε εμά και μηδενική μείωση στις Ηνωμένε Πολιτείε. Γιατί συμβαίνει κάτι τέτοιο. Ένα επιπλέον σημείο είναι να προσπαθήσουμε να δείξουμε στους επενδυτές μας ότι είμαστε αξιόπιστοι εταίροι. Με τους απλήρωτους λογαριασμούς δεν το έχουμε κάνει αυτό ε, πάρα πολλοί ε, δήμαρχοι στη χώρα μου δεν θέλουν να επενδύσουν ιδιαίτερα. Γιατί αν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν θα τους δώσει τα υπεσχημένα, γιατί να αναλάβουν να διατρέξουν κινδύνους. Ένα άλλος τομέας είναι να επιδείξουμε τις βέλτιστες πρακτικές και μάλιστα σε περιπτώσεις όπου μπορεί κανείς να πετύχει στόχους χωρίς βοήθεια από τον κοινοτικό προϋπολογισμό. Πριν 10 χρόνια ήμουν δήμαρχος στην Σλοβακία, 12 χρόνια μάλλον. Και είχαμε στην περιοχή μου, στην πόλη μου, το ταχύτερο ίντερνετ στον κόσμο. Οι καθηγητές επικοινωνούσαν μεταξύ τους ανάμεσα στα σχολεία. Είχαμε επταπλή ταχύτητα βίντεο από τον ισχύοντα τότε κανόνα στην υπόλοιπη Ευρώπη. Και αυτό το κάναμε αποδεικνύοντας ότι οι τοπικές ε, επενδύσεις ε, μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για τον ηλεκτρισμό, για τον καθαρισμό των υδάτων κτλ. Ήταν κάτι το χρήσιμο και αυτό μας επέτρεψε με τα υπόλοιπα χρήματα ε, να μπορέσουμε να βελτιώσουμε το σύστημα επικοινωνίας μέσω του διαδικτύου. Λοιπόν, ε, πρέπει να πάρουμε μέτρα και εκτός αυτών που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σας ευχαριστώ να σας παρακαλέσω επειδή έχουμε να κάνουμε και τις ψηφοφορίες να είστε σύντομοι. Επόμενος είναι ο συνάδελφος. Ε, Έτσι ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα είμαι σύντομος. Θεωρώ ότι η ιδιωτική πρωτοβουλία είναι θέμα ανάληψης κινδύνου. Βλέπω τώρα ότι απλώς είναι ένας τρόπος να αναλαμβάνει κινδύνους που θα καλυφθούν από κάποιον άλλο. Αν υπάρξει λοιπόν κάποια αποτυχία θα πληρωθούν από το δημόσιο τομέα. Εγώ ως πολίτης και αν, υπάρχει ένα πρόβλημα θα πληρώσει ο απλός φορολογούμενος και οι υπεύθυνοι των επιχειρήσεων θα νύψουν τα χείρα τους. Υπήρχε το σχέδιο κάστο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων με την υποστήριξη του Ισπανικού κράτους. Υπήρξε ένα πραγματικό, ένας πραγματικός όλεθρος, γιατί κανείς δεν ανέλαβε τις ευθύνες για αυτά που γινόντουσαν. Τελικά οι Ισπανοί ε, πολίτες πλήρωσαν μερικά δισεκατομμύρια ευρώ από το σχέδιο αυτό που θα πρέπει να τα πληρώνουν επί χρόνια. Το σχέδιο Juncker είναι κάτι το οποίο πρέπει να το αντιμετωπίσουμε με αυτό το πνεύμα ίσως, αλλά θα ήθελα να ρωτήσω την κυρία Γενική Διευθύντρια αν υπάρχει τρόπος να επαναληφθεί το φαινόμενο του σχεδίου Κάστορ με τα προγράμματα τα οποία θα χρηματοδοτηθούν, τα θα από το πρόγραμμα του κυρίου Γιούνκερ και αν τελικά θα μπορέσει να αναλάβει τον κοινό ιδιωτικό τομέα και όχι μονάχα ο δημόσιο προπολογισμό. Μικρό Άλλη, σας ευχαριστώ πολύ συνάδελφοι και αγαπητοί εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας ανακοίνωσε ότι ο προϋπολογισμός του 2015 βασίζεται στις... στο σχέδιο επενδύσεων για την Ευρώπη. Για μας λοιπόν είναι ενδιαφέρον να δούμε πώς θα εξελιχθεί η χρηματοδότηση των επενδύσεων αυτών σε προγράμματα για να υποστηρίξει την πραγματική οικονομία βασιζόμαστε σε μεταβλητά προγράμματα με πραγματική προστιθέμενη αξία για την ευρωπαϊκή κοινωνική οικονομία της αγοράς. Εξ όσων καταλαβαίνω από αυτά που μας λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τα κράτη-μέλη αναμένεται να καταρτήσουν καταλόγους με διάφορα προγράμματα, έργα και μετά μια ομάδα εργασίας ε, που θα είναι υπεύθυνη για την αναθεώρηση των προγραμμάτων να προχωρήσει στην αναθεώρηση λοιπόν των προγραμμάτων των έργων το ερώτημα όμως που ανακύπτει είναι κατά πόσον στέκει η στρατηγική. Η στρατηγική να βασίζεται στον κατάλογο με τις επιθυμίες των κρατών μελών. Γιατί ο κατάλογος με τις επιθυμίες αυτές των κρατών μελών σε διάφορους κλάδους της οικονομίας μπορεί να οδηγήσει σε επικαλύψεις, σε υπέρβαση των οριών ενδεχομένω και έτσι να χάσουμε το δυναμικό του σχεδίου σε ό,τι αφορά την ανάκαμψη της ευρωπαϊκής οικονομίας που αποτελεί και το στόχο. Λαμβάνοντας υπόψη λοιπόν τις ανησυχίες αυτές και ασφαλώς εμείς δεν είμαστε κατά της πρότασης σε καμία περίπτωση να γίνουν προτάσεις από τα κράτη-μέλη. Ωστόσο, οι επενδύσεις θεωρώ ότι θα πρέπει να αποτελούν τμήμα μια ευρύτερης ευρωπαϊκή στρατηγικής η οποία σκοπό θα έχει να καταστήσει ηγετική την Ευρωπαϊκή Ένωση σε πολλούς οικονομικούς κλάδους. Δεν ξέρω αν έχει συζητηθεί αυτό το θέμα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προκειμένου να υπάρξει λίγα πανευρωπαϊκά όμως προγράμματα με σωστή διάρθρωση, προκειμένου να υπάρχει η μέγιστη προστιθέμενη αξία. Τα κράτη-μέλη λοιπόν θα πρέπει να επικεντρώσουν τις προσπάθειές τους ε, σε αυτά ακριβώς τα προγράμματα, και να συμβάλλουν με κάποια συγκεκριμένα στοιχεία τα οποία θα είναι αλληλεοσυμπληρωματικά. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο πρόεδρο, ο επόμενο ομιλητή, ο κύριο Ανώτου. Η ιδέα της μόγλευσης δεν είναι καινούρια, αλλά η κλίμακα στην οποία θα χρησιμοποιηθεί η μόγλευση είναι καινοφανής από, 300, από, 200, από 20 δισεκατομμύρια ευρώ στα 315 είναι μεγάλο, απο, μεγάλο πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα. Η Κομισιόν μιλάει για εγγύηση για προγράμματα υψηλού κινδύνου. Αυτό σημαίνει ότι αν τα προγράμματα αυτά υψηλού κινδύνου τύχουν προτεραιότητας, θα έχουν ένα πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα με μεγαλύτερο από το 15 προς 1. Η δική μου ανησυχία λοιπόν είναι η εξής. Οι επιχειρήσεις θα είναι έτοιμες να αποδηθούν σε αυτό το εγχείρημα. Μήπως απλώς θα είναι ένα πρόγραμμα όπου θα συμμετάσχουν οι επιχειρήσεις, όπου θα υπάρχουν καλές ιδέες, αλλά θα μείνει απ' έξω ο ιδιωτικός τομέας και δεν θα γίνει απολύτως τίποτα. Και τα σχέδια αυτά δεν θα προχωρήσουν. Εγώ φαντάζομαι ότι ο πληθυσμός του Ηνωμένου Βασιλείου έχει βαρεθεί τις ε, συμπράξεις δημόσιου ιδιωτικού τομέα γιατί έχει ήδη αρνητική εμπειρία από τα προγράμματα τα οποία έχουν αναλυθεί στο Ηνωμένο Βασίλειο και τα οποία δεν απέδωσαν καρπούς. Κατανοώ ότι αυτό είναι πολύ διαφορετικό από αυτό το οποίο προτείνεται εδώ για την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά υπάρχει στο Ηνωμένο Βασίλειο μια αρνητική αντίληψη για τέτοιου είδου σχέδια. Γι' αυτό είμαι κάπως σκεπτικιστής σε σχέση με την ικανότητα αυτού του σχεδίου να φτάσει στο επίπεδο των επενδύσεων των 315 δισεκατομμυρίων που λέτε ότι θα πρέπει να προελθούν και από τον ιδιωτικό τομέα. Ευχαριστώ. Ο κύριος Τάραντ είναι ο τελευταίος ομιλητής. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δύο παρατηρήσεις πολύ σύντομα. Καταρχάς να επαναλάβω αυτά τα οποία είπε ο κύριος Λεβαντόφσκι. Ότι αυτές οι εγγυήσεις θα πρέπει να γίνουν ε, ε, ανάμεσα στα δύο ανώτατα όρια των ιδίων πόρων δηλαδή από τη μία και τα ανώτατα όρια των διαθεσίμων από την άλλη. Τώρα για τα χρήματα τα οποία θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν μετά από αποφάσεις των ομάδων υψηλού επίπεδου. Ε, δεν ξέρω τι διαφάνεια μπορεί να υπάρξει, δεν ξέρω πώς ακριβώς το βλέπει να το κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η ομάδα αυτή υψηλού επίπεδου θα ασχοληθεί και με επενδυτικά γενικά προγράμματα και κυρίως με προγράμματα στον τομέα των υποδομών. Ε, εμείς θα πρέπει να γνωρίζουμε ποιοι θα αποτελέσουν την ομάδα αυτή ποιοι θα οριστούν στην ομάδα αυτή και ο ορισμός θα πρέπει να γίνει και με τη δική μας συνεργασία γιατί αλλιώς θα καταλάβουμε, θα καταλήξουμε μάλλον σε μια άλλη ομάδα υψηλού επίπεδου ε, την σχετική με την ρύθμιση των φορολογικών θεμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ήταν συναντήσεις στις οποίες συμμετείχαν μεγάλες λογιστικές εταιρείες όπως η KPMG και η Price Waterhouse. Γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα να μην κάνει καμία σύσταση ομάδας η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χωρίς την δική μας συνένεση. Υπάρχουν και άλλοι ομιλητές, αλλά έχουμε κλείσει τον κατάλογο των ε, αγορεύσεων. Κυρία Γενική Διευθύντρια, έχετε ακούσει τις ανησυχίες και τις ερωτήσεις των βουλευτών μας. Σας παρακαλώ να είσαστε σύντομοι. Έχουμε κάθε κατανόηση για το γεγονός ότι δεν μπορείτε να απαντήσετε όλα τα ερωτήματα. Η Κομισιόν ξέρω ότι πρέπει να σκεφτεί για να μπορέσει να απαντήσει πολλά από αυτά τα ερωτήματα. Είμαστε έτοιμοι να δεχτούμε απαντήσεις γραπτός αν μπορείτε να μας ε, υποσχεθείτε ότι μπορείτε να απαντήσετε γραπτός μέχρι την επόμενη συνεδρίασή μας, νομίζω θα έχουμε πολύ καλύτερο έδαφος για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε το θέμα αυτό και έτσι στην επόμενη συνεδρίασή μας θα μπορέσουμε να το συζητήσουμε καλύτερα. Σας παρακαλώ λοιπόν να απαντήσετε για τα κομμάτια τουλάχιστον μπορείτε εσείς να απαντήσετε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε να απαντήσω σε τμήματα των ερωτήσεων και φυσικά θα είμαστε ε, σε διαρκή επαφή και μπορούμε και γραπτά να απαντήσουμε στις ερωτήσεις σας. Και προφανώς ε, οι λεπτομέρειες θα πρέπει να διαμορφωθούν στην πορεία. Είναι δύσκολο να είμαστε λίγο πιο σαφείς πριν τον Γενάρη. Φυσικά είναι λίγες οι εβδομάδες που μας χωρίζουν από τον Γενάρη για να απαντήσω όμως σε κάποια από τα ερωτήματα των αξιότιμων βουλευτών. Για τη μόχλευση αρχικά και πώς δουλεύει η μόχλευση. Η εκτίμησή μας είναι ότι δεν υπάρχει έλλειψη πόρων ρευστότητα ή αποταμιεύσεων στην Ευρώπη. Θεωρούμε ότι οι αποταμιεύσει είναι σε ιστορικά υψηλό επίπεδο, αλλά οι επενδύσει παρόλα αυτά δεν κινητοποιούνται, δεν διοχετεύονται στην πραγματική οικονομία. Γιατί υπάρχει μεγάλη, ε, μεγάλος φόβος για τον κίνδυνο, για το ρίσκο και αυτό είναι γεγονός. Γι' αυτό λοιπόν πιστεύουμε ότι ο ευρωπαϊκός Προπολογισμό μπορεί να χρησιμοποιηθεί καλύτερα αν αντί να επικεντρωθεί στις επιδοτήσεις μπορεί να εκμεταλλευτεί την τρέχουσα κατάσταση των χρηματοπιστωτικών αγορών και να επωφεληθεί από τη μόχλευση αυτή. Όπως σας εξήγησα λοιπόν, αυτή η ανάλυση κινείται σε δύο επίπεδα. Καταρχάς, η ο δανεισμός της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων στην αγορά και μετά η συμμετοχή στα προγράμματα. Αυτό μας οδηγεί στο συντελεστή 15, 15 ως μόχλευση. Και αυτό είναι μια συντηρητική εκτίμηση, να σας πω την αλήθεια. Αυτό κάποιοι μπορεί να το θεωρήσουν χρηματοοικονομικό ε, μηχανικό τρόπο. Εμείς θεωρούμε ότι αποτελεί τον καλύτερο τρόπο αξιοποίησης των χρημάτων. Κάτι άλλο τώρα για τον κίνδυνο. Πώς αντιμετωπίζουμε το ρίσκο. Θέλουμε να συμπληρώσουμε τα προγράμματα τα οποία ήδη υφίστανται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στον Ευρωπαϊκό Προϋπολογισμό και στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων προκειμένου να αναλάβουμε δραστηριότητες με μεγαλύτερο ρίσκο σε ό,τι αφορά το μακροπρόθεσμο ότι η μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση των προγραμμάτων είναι διαφορετικά φυσικά τα πράγματα αυτά σε ό,τι αφορά και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Να δούμε λοιπόν πώς θα αντιμετωπίσουμε τους διαφορετικούς αυτούς κινδύνους. Αλλά αυτό το κίνδυνο θέλουμε να στοχεύσουμε και γι' αυτό λοιπόν πιστεύουμε και θέλουμε να υπάρχει μια καλά χρηματοδοτούμενη εγγύηση 15%. Ένα τρίτο ζήτημα που ακούσαμε είναι ποιος θα είναι ο αντίκτυπος στον προπολογισμό του 2015. Θα σας δώσουμε λεπτομέρειες για το σχέδιο πληρωμών σε ό,τι αφορά και τις συμβολές μας για το Ταμείο Εγγύησεων. Φυσικά οι εγγυήσει θα πρέπει να φτάσουν και πέρα από το 2020, γιατί μιλάμε για μακροπρόθεσμες χρηματοδοτήσεις. Δεν πρόκειται για ένα πρόγραμμα το οποίο θα ολοκληρωθεί στο τρέχον πολίτες δημοσιονομικό πλαίσιο. Αλλά το 2015 δεν υπάρχει ανάγκη επιπρόσθετων πληρωμών. Θα υπάρξει όμως αναδιανομή των ε, πιστώσεων για το Connecting Europe και για το Horizon 2020 από τη σχετική γραμμή του προπολογισμού. Αυτό το είπα και προηγουμένω. Σε ό,τι αφορά το πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο, δεν πιστεύουμε ότι θα πρέπει να το υπερβούμε. Το πρόγραμμα λοιπόν θεωρούμε ότι μπορεί να καλευτεί στα πλαίσια και στα περιθώρια του πολιτικού δημοσιονομικού πλαίσιο, στα ετήσια περιθώρια καταρχάς και κατά δεύτερον στο συνολικό ε, περιθώριο δεσμεύσεων που όπως ξέρετε σκοπό έχει την ανάπτυξη, ιδιαίτερως για τη νέα και για την, για ε, την νεολαία και για την ανάπτυξη. Σε αυτό θα στοχεύσουν άλλωστε και οι πρωτοβουλίες που θα υποβάλουμε για τις συμβολές των κρατών μελών. Θα σημειώσατε ότι ήδη στη δημόσια ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής υπάρχει αναφορά σε ενδεχόμενη ε, ιδιαίτερη μεταχείριση στα πλαίσια του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης σε ό,τι αφορά τις ε, εθνικές συνεισφορές στο Ταμείο. Γιατί προφανώς ένα τμήμα μπορεί να γίνει σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά και τα κράτη-μέλη και το εθνικό επίπεδο πρέπει να είναι σημαντικό. Και γι' αυτό λοιπόν στο επόμενο Συμβούλιο της επόμενης εβδομάδας θέλουμε δέσμευση από τα κρατη για να διπλασιάσουν τα χρηματοοικονομικά μέσα στα πλαίσια του Ταμείου. Για να απαντήσω λοιπόν σε κάποια ερώτηση, υπάρχει έκκληση ουσιαστικά για πιο αποτελεσματική χρήση των χρηματοοικονομικών μέσων που δεν έχουν αξιοποιηθεί στο βαθμό το βέλτιστο θεωρούμε. Και τέλος, συμφωνώ με τον βουλευτή που ζήτησε να υπάρξει όσο πιο απλή διαμόρφωση γίνεται. Γιατί τελικά όταν ξεκινούν διαπραγματεύσει, σε πολλέ περιπτώσει καταλήγουμε με σενάρια και προγράμματα τα οποία είναι πάρα πολύ δύσκολο να εφαρμοστούν στην πράξη. Άρα, η δική μα προσέγγιση είναι η εξή. Όσο σημαντικά είναι τα χρήματα και οι εγγύησει, είναι και το να υπάρξει ένα καλό πλαίσιο για επενδύσεις, καλύτερη ρύθμιση, κατάργηση των εμποδίων στις επενδύσεις. Σε αυτό θα καταναλώσουμε πολύ μεγάλο τμήμα της ενεργειάς μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ερωτήσεις που μου θέσατε και προφανώς ε, ευχαρίστως θα συνεχίσουμε να σας απαντάμε και γραπτά στις ερωτήσεις. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο Πρόεδρος. Σας ευχαριστώ λέει και ο Πρόεδρος. Δεν θα κάνω περαιτέρω σχόλια. και βέβαια θα πρέπει να επανέλθει η Κομισιόν στα συγκεκριμένα ερωτήματα. Σας ευχαριστώ για τη συζήτηση, για την ε, παρέμβαση της Κομισιόν. Περνάμε στο επόμενο σημείο και τώρα είναι η γνωμοδότηση του κυρίου Τάραντ για την έκθεση του, της υπάτη, υπάτης εκπροσώπου για τα θέματα εξωτερικής πολιτικής. Κύριε Τάραντ, τηλεγραφικά αν μπορείτε. Σας ευχαριστώ. 30 δευτερόλεπτα κύριε Πρόεδρε. Είναι μια ακόμα περίπτωση όπου η Επιτροπή, Εξωτερικών Υποθε... η Επιτροπή Προϋπολογισμών προσπαθεί να χώσει τη μύτη στα χωράφια άλλων επιτροπών και να συστήσουμε σε άλλες επιτροπές πώς να χρησιμοποιήσουν τους ε, πόρους τους. Πρέπει να πω και εδώ ότι το πρόβλημα των πληρωμών είναι πάλι ένα πάρα πολύ κεφαλαιόδες πρόβλημα που πρέπει να αντιμετωπίσουν τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα επανέλθουμε τον Ιανουάριο Όλοι θέλουν να ψηφίσουν όμως και ίσως πρέπει να περάσουμε στις ψηφοφορίες τώρα. Ωραία, πολύ ωραία, πολύ σύντομα. Ήμουν έτοιμος να κρατήσω, να χρόνο με το χρονόμετρο, αλλά αφαιρέθηκα. Ερχόμαστε λοιπόν στις ψηφοφορίες. Δεν ξέρω αν μπορεί και η ομάδα μου να με βοηθήσει να ξέρω τι πρέπει να ψηφίσω. Όχι, δεν θέλω τον κατάλογο ψηφοφορίας του ΕΛΚ. Σας ευχαριστώ. Δεν θα πάρω. Ξεκινάμε. Με, τον, με την ε, έκθεση Ντεπρές και Λεβαντόφσκι που ήταν αντικείμενο συζήτησης πριν από λίγο. Τροπολογία 1 του εισηγητή που φυσικά την υποστηρίζει. Ψήφι υπέρ. Κατά. Κανεί Α, εγκρίνεται. Τροπολογία 2. Του εισηγητή, των εισηγητών εισηγητές είναι υπέρ. Ποιος είναι υπέρ. Όλοι. κανεί κανείς, κατά. Εγκρίνεται. Παράφος 4, τροπολογία 14 των εισηγητών κατά αποχές, μία αποχή, μία ψήφος κατά, μία αποχές, όχι εγκρίνεται. Τροπολογία 15. Οι εισηγητές είναι κατά. Α, εκπίπτει, εκπίπτει γιατί εγκρίθηκε η 14, σωστά. 16 οι ίδιοι ε, συντάκτες, οι συζητητές είναι κατά ψήφι υπέρ. Ο συντάκτης και δύο, τρεις, ποιοι είναι κατά, οι υπόλοιποι σχεδόν, απολύπτεται. 17 έχει αποσυρθεί, τροπολογία 4, ο εισηγητής την υποστηρίζει, ψήφι υπέρ. Πολύ. Κατά. Λίγοι. Τέσσερις. Αποχές. Κανείς. Εγκρίνεται. Τροπολογία 5. Αιτιολογική σκέψη Β. Έχει αποσυρθεί. Η τρία παίζει ακόμα. Δεν πρέπει να την ψηφίσουμε. Όχι, όχι. Την 6. Την 6. Ψηφίσουμε. Οι εισηγητές είναι εναντίον εδώ. Ποιος υποστηρίζει την έξι τώρα. Κανείς. Κατά. Όλοι. Απορρίπτεται. Τροπολογία επτά των εισηγητών. Υπέρ. Προφανώς. Είναι οι εισηγητές. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Μία ψηφός κατά. Δύο ψήφοι κατά. Δεν, δεν είδα αν ψηφίσετε υπέρ ή όχι. Α, εντάξει, υπέρ. Μία ψήφος κατά τελικά, αποχές. Καμία αποχή εγκρίνεται. Η 8 εκπίπτει. <clears throat> Μάλλον καλύπτεται την 7. Ερχόμαστε σε μία προφορική τροποποίηση του εισηγητή για την αιτιολογική σκέψη Δέλτα. Οι εισηγητέ είναι προφανώς υπέρ, ψήφι υπέρ. πολύ, κατά, κανείς, αποχές, ε, ένα άτομο κατά μάλιστα. Αποχές, εγκρίνεται με μία ψηφομονάχα κατά, τροπολογία 9, για την ίδια διαλογική σκέψη, ψήφι κατά, περισσότεροι, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 10 έχει αποσυρθεί όμως. Τροπολογία 11 των εισηγητών, η οποία είναι υπέρ. Φυσικά ποιος είναι υπέρ. Κατά. 2. αποχέ, Αποχές. Εγκρίνεται. Χωρίς αποχές. Τροπολογία 12. Πάλι των εισηγητών. Υπέρ. Ευχαριστώ. Κατά. Μία ψήφος κατά. Αποχές. Καμία εγκρίνεται. Τέλος η τροπολογία Moody 13. Οι συγητές είναι κατά. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονικός έλεγχος. Δύο δεν έχουν ψηφίσει ακόμα. τρει δεν έχουν ψηφίσει. Κάποιο βρήκε την κάρτα του όμως. Έχουμε 29 ψήφου που καταγράφηκαν, κλείνω την ε, ψηφοφορία 14 υπέρ, 13 κατά, 2 αποχέ. με μικρή πλειοψηφία, αλλά εγκρίνεται. Τελική, ψηφο... τελική ψηφοφορία, ηλεκτρονικά βέβαια. Άρχεται η ηλεκτρονική ψηφοφορία. Εντάξει. πέρας της ψηφοφορίας. 30 υπέρ, μία ψήφος κατά, καμία αποχή. Ευχαριστώ πολύ. Συγχαρητήρια στους εισηγητές μας. Και περνάμε λοιπόν τώρα στην έκθεση της κυρίας Βάνα που είμαι εγώ σκιώδης εισηγητής. Πρόκειται για ένα έργο στην Ελλάδα για το Ευρωπαϊκό Τομείο προσαρμογή στην παγκοσμιοποίηση. Κύρκος 1 ε, υπέρ, η τροπολογία είναι υπέρ. Κατά. Κύρτσος, συγγνώμη. Τρει κατά. Αποχές. Κανείς εγκρίνεται. Δεύτερη τροπολογία δική μου και η σύγκριτρια είναι υπέρ. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 3. Ούλσκο και Λυπή από την Επιτροπή Απασχόλησης. Η συγκήτρια είναι υπέρ. Ποιος είναι υπέρ? Κατά. Κανείς. Αποχές. Κανείς. Έγκρινεται. Η ίδια η συγκήτρια και η συγκήτρια είναι υπέρ. Ποιος την ακολουθεί, ποιος είναι υπέρ. Κατά. Κανείς, αποχές, εγκρίνεται. Πέντε, του κυρίου Κίρτσου. Ε, συν, πρόσημο, υπέρ. Κατά. Ένας. Αποχές. Εγκρίνεται. Η έξι. Επιτροπή Επασχόλησης. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Ομοφωνία. 7. ίδια εισηγήτρια. Θετικό πρόσημο υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. 8. ίδια διαδικασία. Ποιος είναι υπέρ παρακαλώ. Κατά. Κανείς. Άποχες. Εγκρίνεται. Η 9. Επίσης από την Επιτροπή Επασχόλησης υπέρ. Κατά. αποχές τελική ψηφοφορία ηλεκτρονικά. Τώρα λοιπόν ψήφισαν όλοι. υπέρ ψηφοφορίας 28 υπέρ 2 κατά εγκρίνεται. Και τώρα περνάμε και πάλι από το Ταμείο της ε, Παγκοσμιοποίησης στην έκθεση Τσάνι. Να ξεκινήσουμε με την τροπολογία 2 για την παράγραφο 1 από την Επιτροπή Απασχόλησης. Κατά ο εισηγητής υπέρ. Δεν κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Η τρία της Επιτροπής Απασχόλησης με την ίδια διαδικασία, η κατά ο εισηγητής. Ποιος είναι υπέρ της τροπολογίας. Η πράσινη και η ελεύθερη και το ECR. Κατά. Οι χριστιανοδημοκράτες και οι σοσιαλιστές, πλειοψηφία, ποιος απέχει. Απορρίπτεται. Η τέσσερα και πάλι της Επιτροπής Απασχόλησης, η διαδικασία παρακαλώ. Υπέρ. Κατά. Και κρυφά κρυφά η κυρία Χόλμαγερ. Και κατά οι υπόλοιποι. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική α του εισηγητή που συμπληρώνει τις τροπολογίες 5 και 6 και είναι υπέρ. Ο εισηγητές ποιος είναι υπέρ. Όλοι κατά. Κανείς εγκρίνεται και περνάμε λοιπόν στην 7 Ποιο είναι υπέρ. Θετικό πρόσημο έχει βάλει ο Συγητή. Κατά. Οι χριστιανοδημοκράτε δεν φτάνουν όμω, ποιο απέχει. Εγκρίνεται η 8 της Επιτροπής Απασχόλησης. Αρνητικό πρόσημο έχει βάλει ο συγητής. Ποιος είναι υπέρ της τροπολογίας της Επιτροπής Απασχόλησης Πράσινη, Φιλεύθερη. Ποιος είναι κατά. Όλοι οι υπόλοιποι Απορρίπτεται. Τροπολογία 9. Και πάλι της Επιτροπής Απασχόλησης η διαδικασία κατά ο εισηγητής ή ποιος είναι υπέρ της Επιτροπής της Τροπολογίας 9. Δεν φτάνουν. Κατά. Πολύ. Ποιος απέχει. Απορρίπτεται η 10 επίσης της Επιτροπής Απασχόλησης. Ο εισηγητής είναι κατά. Ποιος ε, είναι υπέρ. οι σοσιαλδημοκράτες, οι φιλελεύθεροι, οι πράσινοι και οι αριστεροί. Ποιος είναι κατά. Οι λίγοι υπόλοιποι χριστιανοδημοκράτες και το EFTD. Αποχές. Νομίζω πλειοψηφία είναι κατά. Του κύριου Ντενανό ή... Α, συγγνώμη λέει ο Πρόεδρος. Ποιος είναι υπέρ της ε, τροπολογίας της Επιτροπής Επασχόλησης. Τη 10, τη 10 να την ψηφίσουμε ηλεκτρονικά για να έχουμε καλύτερη εντύπωση, λέει ο Πρόεδρος. Στη 10, στη 10 έχουμε φτάσει. Τροπολογία 10, στην παράγραφο 7D. Ναι, συγγνώμη, σας μπέρδεψα λίγο. Να δούμε, να δούμε τι κάνουν οι χριστιανοί κύριε Πρέντα. Λείπει μία ψήφο. Ψήφισατε όλοι. Ε, κάποιος δεν θέλει. Πέρας ψηφοφορίας. 19 υπέρ. 8 κατά. Εγκρίνεται η τροπολογία 10. Πάμε στην 11 του κύριου Ντένανο για την παράγραφο 8. Ποιος είναι υπέρ. Όλοι. Κατά. Το Ισιάρ. Αποχές. Είναι πράσινη εγκρίνεται η 12 της Επιτροπής Απασχόλησης. Θετική σύσταση του Επιτροπή. Ποιος ακολουθεί τον, ε, τον εισηγητή. Κατά. Κανείς. Αποχές. Εγκρίνεται η 13 πάλι της Επιτροπής Απασχόλησης κατά ο εισηγητής. Ποιος θέλει να υπερψηφίσει την τροπολογία 13 της Επιτροπής Απασχόλησης. Η αριστερή κατά πολύ. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 1. Δεν ε, συστήνει ο εισηγητής. Ποιος είναι υπέρ. Ο εισηγητής, ναι. Και φιλελεύθερη. Όχι. Δύο υπέρ, κατά. Όλοι οι υπόλοιποι απορρίπτεται και περνάμε στην τελική ψηφοφορία ηλεκτρονικά παρακαλώ. Dann ist die Abstimmung geschlossen. Εγκρίνεται με μία μόνο ψήφο κατά συγχαρητήρια κύριε Τσάνη. Ερχόμαστε σε μία άλλη έκθεση για το Ταμείο παγκοσμιοποίηση. Είναι η έκθεση του κυρίου Όλμπρεχτ για την Fiat στην Πολωνία. Τροπολογία 1. Ο είναι υπέρ, ψήφι υπέρ. Πολύ κατά, κανείς, αποχές, εγκρίνεται ομόφωνα. Τροπολογία 2 του εισηγητή είναι υπέρ, ψήφι υπέρ, κατά, αποχές, ομόφωνα. Τροπολογία 3 πάλι του εισηγητή που την υποστηρίζει υπέρ, κατά, αποχές, ομόφωνα. Τροπολογία 4 και πάλι του εισηγητή υπέρ κατά άποχες ομόφωνα. Τροπολογία 5 την υποστηρίζει ο εισηγητής. Ψήφι υπέρ κατά άποχες μία αποχή εγκρίνεται. Τροπολογία 6 πάλι την υποστηρίζει ο εισηγητής. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται ομόφωνα και 7 πάλι της Επιτροπής Απασχόλησης υποστηριζόμενη από τον εισηγητή ψήφι υπέρ κατά αποχές μία εγκρίνεται τελική ψηφοφορία ηλεκτρικά. Λείπει μία ψήφος. Δεν θέλει να ψηφίσει. Εντάξει, κλείνουμε την ε, ψηφοφορία. 27 ψήφοι υπέρ, μία κατά, καμία αποχή. Συγχαρητήρια στον κύριο Όλμπρεχτ. Περνάμε στο επόμενο θέμα. Πάλι από το Ταμείο Παγκοσμιοποίηση για την Whirlpool. Μπορούμε να ψηφίσουμε όλε τι τροπολογίε από κοινού αν συμφωνείτε. Του κυρίου Βιώτη, ο εισηγητή θέλει να εγκριθούν όλε. Μόνο την τελευταία αμφισβητούν οι χριστιανοδημοκράτες. Μπορούμε να ψηφίσουμε την 1 μέχρι την 9 όλε μαζί. Ο κύριο Βιώτη τι υποστηρίζει. Ποιοι υποστηρίζουν την έγκριση της 1 μέχρι 9. Πολύ κατά αποχές κανείς ομόφωνα ή 1 με εγκρίθηκαν. Πάμε στην 10. Ο εισηγητής είναι υπέρ. Ποιο είναι υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονικά θα το ελέγξουμε. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. 13-14 απορρίπτεται με δύο αποχές. Τελική ψηφοφορία ηλεκτρονικά. Άρχεται. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται με μία ψηφοκατά και χωρίς καμία αποχή. Συγχαρητήρια κύριε Βιώτη. Μεταφορές. μεταφορές. Μου λέει η γραμματεία ότι 40, 46, 49, 50 και 55 είναι αυτές που έχουμε εγκρίνει ήδη σε πολιτικό επίπεδο. Είναι συνέπειες για τον προϋπολογισμό αυτών που έχουμε εγκρίνει ήδη προηγουμένως. Θεωρώ λοιπόν ότι υπάρχει μια πλειοψηφία. Σας προτείνω να τις ψηφίσουμε unblock όλες μαζί. Αν δεν υπάρχει αντίρρηση λοιπόν ψηφίσουμε όλες μαζί ποιος είναι υπέρ αυτών. Κατά. Μία ψήφος κατά. Αποχές. Καν μία. Δύο. Μία ψήφος κατά και μία αποχή. Εγκρίνονται λοιπόν. Περνάμε στην 55 για το κτίριο Jean Monnet. Στο σημείο 15 μάλλον, συγγνώμη. Θέλει να πει κάτι η κυρία Χολμάιερ. Την τελευταία φορά ενημέρωσα ότι το να υπάρχει διαφορετικά, ε, διαφορετική, διαφορετικά γραφεία για το προσωπικό είναι πολύ δύσκολο σε ό,τι αφορά τα επιπλέον έξοδα και τα 20 εκατομμύρια που θα πρέπει να μεταφερθούν μέχρι το επόμενο χρόνο. Μάλιστα, λέει ο Πρόεδρος. Το κοιτάξαμε αυτό. Ποιο θέλει να ε, εγκρίνει αυτή τη μεταφορά 55. Όλοι. Ή κατά. Κανείς. Κανείς ε, θέλει να απόσχει. Μία αποχή. Με μία αποχή λοιπόν σχεδόν ομόφωνα λάβαμε την απόφαση αυτή και περνάμε στον προπολογισμό 2014 στις λοιπές, στα λοιπά τμήματα και πάλι για μεταφορές πρόκειται τις οποίες πρέπει να ψηφίσουμε μία-μία. Μόνικα, μπορεί να ψηφίσουμε όλους μαζί. Τα έχουμε κοιτάξει από το προηγουμένο τα θέματα αυτά. Είναι κανείς κατά της ε, ψηφοφορίας ο κύριος Δεπρέ. Δεν είναι αντίρρηση, κύριε Πρόεδρε. Βλέπω ότι πρόκειται για την αγορά της οικίας του εκπροσωπού της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Αλβανία για περίπου 1,5 εκατομμύριο. Δεν είμαι γνώστης των αλβανικών οικοδομικών δεδομένων. Δεν ξέρω αν είναι οι ίδιες τιμές όπως τις άλλες μεγάλες πρωτεύουσες της ε, Ευρώπης. Δεν ξέρω λοιπόν αν ένα μέγαρο, πολλά μέγαρα ή μία παράγκα. Μου φαίνεται κάπως υψηλό το ποσό. Σα ευχαριστώ. Ναι, είναι σαφέ και εγώ παρόμοια ερωτήματα είχα όπω και εσείς κύριε Ντεπρέ. Το ερώτημα αυτό το ξέρω από τις πρεσβείες, όπου οι οικίες των πρεσβευτών δεν είναι μόνο οικίες και κατοικίες, αλλά και μία έντρα. Αλλά όντως 1,6 εκατομμύρια στην Αλβανία αναρωτιόμαστε τι αγοράσαμε. Και μήπως η διαδικασία αυτή δεν ξέρω αν είναι φυσιολογική και η λαμβανική αντιπροσωπεία ε, θα είναι πιο κανονική στη λειτουργία της πλέον ή μήπως αυτό πραγματικά είναι περίεργο. Εδώ έχουμε λοιπόν να διευκρινίσουμε κάποια ερωτήματα. Η Μόνικα, ναι, καταρχάς ε, τα έλαβα αυτά τελευταία στιγμή, αλλά θεωρώ ότι θα λάβουμε μία κοινοποίηση και ότι πρόκειται μόνο για προσωρινή μεταφορά προκειμένου μέχρι το Μάρτιο να έχουμε τη σχετική κοινοποίηση, γιατί ως τώρα δεν έχουμε σχετική κοινοποίηση για κτίριο στην Αλβανία. Γι' αυτό όλοι προτείνω να κάνουμε τη μεταφορά, αλλά υπό τον όρο να λάβουμε συγκεκριμένες και ακριβεί πληροφορίε προτού δαπανηθούν τα χρήματα αυτά και προτού απελευθερωθούν τα κονδύλια αυτή. Να γίνει μεταφορά λοιπόν ε, στα τέλη του χρόνου μέχρι το επόμενο έτος και μέχρι το Μάρτιο να λάβουμε πληροφορίες. Όχι οριστική λοιπόν έγκριση, αλλά μία μεταφορά μέχρι να λάβουμε ακριβείς πληροφορίες για αυτό το κτίριο στα Τυρανα. Και μετά να αποφασίσουμε αν το αγκρίνουμε. Μάλιστα, χρήσιμες πληροφορίες λέει ο Πρόεδρος, δηλαδή μεταφέρουμε τα κονδύλια αυτά στο επόμενο έτος. Κύριε Ντεπρέ, θέλετε πάρει το λόγο. Συμφωνώ, λέει κύριος Ντεπρέ. Λοιπόν, Έχουμε τέσσερις μεταφορές. Ρώτησα αν μπορούμε να τις ψηφίσουμε όλες μαζί. Συμφωνεί, συμφωνούμε λοιπόν με αυτά τα οποία είπε η κυρία Χολμάρ. Δεν αγοράζουμε το κτίριο, απλώ κάνουμε τη μεταφορά στον προπολογισμό 2015. Μπορούμε να τα ψηφίσουμε λοιπόν όλα αυτά τα τέσσερα αιτήματα μεταφορά. Ψήφι υπέρ παρακαλώ. Κατά. Τέσσερι. Αποχέ. Δύο. Έχουν αποφασιστεί λοιπόν και αυτές τις μεταφορές. Ένα ακόμα σημείο για την πολιτική κτηρίων. Ήδη νομίζω ότι την τελευταία φορά είχαμε, ήμασταν έτοιμοι να το εγκρίνουμε αλλά δεν το έχουμε κάνει ακόμα. Είναι ο χώρος επισκέψεων, επισκεπτών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις Βρυξέλλες. Θέλετε να το συζητήσουμε. Όχι. Μπορούμε να ψηφίσουμε, να αποφασίσουμε. Ναι. Ποιος είναι υπέρ. Ευχαριστώ. Κατά. Τέσσερις ψήφι κατά. Αποχές. Μία. Εγκρίνεται λοιπόν και αυτή η μεταφορά. Τελειώσαμε λοιπόν τις ε, ψηφοφορίες. Υπάρχει κάτι στα διάφορα. Παρατηρήσεις. Όχι. Πέραση συνεδριάσεω, συνεδριάσεως θα τα πούμε στο Στρασβούργο.